Okay, colleagues. I think um, I know there's a lot to catch up on after summer holiday. Καλημέρα σας. Για να ξεκινήσουμε, έχουμε πολλές εκκρεμότητες γιατί έχουμε διακόψει και για το καλοκαίρι. Θα ήθελα λοιπόν να σας παρακαλέσω να καθίσετε. Είναι ήδη 9 και 4 και έχουμε προσκεκλημένους θα ήθελα λοιπόν να ξεκινήσουμε όσο το δυνατόν πιο πολύ στην ώρα μας. Ελπίζω όλοι να περάσατε καλά, να ξεκουραστήκατε το καλοκαίρι και να έχετε επιστρέψει έτοιμοι για σκληρή προσπάθεια τους επόμενου μήνες και μέχρι ε, τις ε, την επόμενη διακοπή για τα Χριστούγεννα πολύ βαρύ το πρόγραμμα σήμερα το πρωί, αλλά και για την επόμενη ε, μια μισή ημέρα. Θα ξεκινήσω λοιπόν με την έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Θα ήθελα να μου πείτε, εγκρίνετε. Έχετε κάποιες ε, ή αλλαγές που να επιθυμείτε. Όχι, εγκρίνετε. Δεύτερον, έχουμε τις ανακοινώσεις Προεδρίας. Πρώτα απ' όλα για την επόμενη εβδομάδα, 6 Σεπτεμβρίου το απόγευμα, για μια φορά ακόμα το Κοινοβούλιο θα φιλοξενήσει τους ε, πρέσβεις και τους επικεφαλείς των αντιπροσωπιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σίγουρα έχετε λάβει πρόσκληση για μια σειρά εκδηλώσεων την επόμενη Τρίτη. Η πρώτη είναι στις 3 που είναι η εναρκτήριο συνεδρίαση για τον τρόπο που μπορούμε να επικοινωνήσουμε την Ευρώπη σε τρίτες χώρες και μετά έχουμε τρία παράλληλα σεμινάρια από τις 3 και 4 μέχρι τις 4 και 45 και μετά πάλι στις 5 θα έρθει ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου, ο κύριος Σούλς, όπως επίσης και η κυρία Μογκερίνη, για να συζητήσουν με τους επικεφαλείς των αντιπροσωπείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στο εξωτερικό. Είναι μια σημαντική δυνατότητα να συναντηθείτε με τους πρέσβεις και αν σας ενδιαφέρει κάποια συγκεκριμένη χώρα, πολλές φορές μπορείτε να έρθετε και σε επαφή ε, με το άτομα που γνωρίζει καλύτερα ποια είναι τα θέματα που τους απασχολούν στις αντιπροσωπείς τους και υπάρχουν ε, διάφορα θέματα, όπως για παράδειγμα τα 3.000 άτομα τα οποία περισυλλέγησαν χτες στα ύδατα ε, της Λιβύης από διάφορα ευρωκά σκάφη. Ξέρετε πως εκεί έχουν ενταθεί οι προσπάθειες διάπλου και έχουμε και την ανθρωπιστική κρίση στη Συρία που όλο και χειροτερεύει. Σας παρακαλώ λοιπόν την επόμενη Τρίτη ελάτε να συναντηθείτε με τους πρέσβεις. Στις 27 Σεπτεμβρίου από τις 9 και μέχρι τις 11 θα γίνει μια έκτακτη συνάντηση της Επιτροπής μας έτσι ώστε να ανταλλάξουμε απόψη με τον, με τον Επίτροπο Μίμητσα για την Ευρωπαϊκή Συνένωση, Συνένεση με για την ανάπτυξη. Το μεγάλο θέμα που έχουμε μέχρι και τα Χριστούγεννα, σημειώστε το στην ατζέντα σας, 27 Σεπτεμβρίου, ημέρα Τρίτη, 9 το πρωί με 11. Θα ήθελα να σας ανακοινώσω πως και για το θέμα του σημείου 4 θα έρθει να μας δει ο, ο Γενικός Γραμματέας για θέματα ΑΚΕ ε, και θα συζητήσουμε το, την επόμενη εποχή ε, στην πλαίσια της Συμφωνίας Κοτονού, οπότε περιμένουμε να συζητήσουμε τα θέματα αυτά μαζί του. Τώρα για τις ανακοινώσεις δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να θέσετε, όχι. Περνάμε λοιπόν στο σημείο 3 που είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι ανακοινώσει Τώρα μόλις τελείωσε το καλοκαίρι Ξέρω όμω πως έχουμε νέο συνάδελφο την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον Κάρστεν Σόρενσον, που πρόκειται να μα συστηθεί γιατί έχει ε, αντικαταστήσει την Κάθριν. Σα ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Δεν έχουμε κάποιες ιδιαίτερε ανακοινώσει για το περιεχόμενο. Θα ήθελα να χρησιμοποιήσω την ευκαιρία αυτή και να σας συστηθώ. Είμαι στην DG DEFCO, στην ε, μονάδα για τις ε, ε, σχέσεις με τα υπόλοιπα όργανα και είμαι αναπληρωτής επικεφαλής μονάδας αυτής. Χαίρομαι λοιπόν που θα έχω την ευκαιρία να συνεργαστώ μαζί σας. Και εμείς σας καλωσορίζουμε και θα συνεργαστούμε μαζί σας εξίσου καλά, όπως και με την προκάτοχό σας. Ξέρω πως υπάρχουν πολλά θέματα, έχουμε τη συνένεση για την ανάπτυξη, τη Συμφωνία Κοτονού κτλ. Μπορούμε να περάσουμε στο 4 που είναι το βασικό σημείο που είναι η αξιολόγηση της εταιρικής συμφωνίας με το Κοτονού. Θα ακούσουμε τι ε, θα μας πει ο Νόρμπετ Νόιζερ για τις σχέσεις μετά το 2020. Πριν όμως κάνουμε κάτι τέτοιο, με μεγάλη χαρά να καλωσορίσουμε τον Κουν Ντούνς, που είναι διευθυντής στην Γενική Διεύθυνση ΔΕΦΚΟ και ο οποίος θα μας μιλήσει σήμερα για μια αξιολόγηση που έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η ΥΠΑΤΗ Αρμοστής για την συμφωνία αυτή του Κοτονού. Είναι λοιπόν μια ευκαιρία για να ακούσουμε ποια είναι τα αποτελέσματα της αξιολόγησης από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να κάνουμε και τις ερωτήσεις που χρειάζεται. Κύριε Ντούνς, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Είναι μεγάλη χαρά που μπορώ και εγώ να ξεκινήσω ε, τη χρονιά μετά το καλοκαίρι, μιλώντας για ένα τέτοιο θέμα, είμαι διευθυντής στη Γενική Διεύθυνση ΔΕΦΚΟ και είμαι διευθυντής για τα θέματα της σχέσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση, για την Νότια Αφρική, ε, γεωγραφικά την η Ανατολική Αφρική, όπου επίσης και για τη Task Force για τα θέματα με τη συμφωνία με του Κουτουνού με την, ε, στα πλαίσια της Γενικής Διευθυνσής ΔΕΦΚΟ και θα ήθελα σήμερα να σας παρουσιάσω την αξιολόγηση την οποία μόλις ε, φέραμε σε πέρας. Η αξιολόγηση αυτή έγινε σε συνεργασία και με άλλους ε, συναδέλφους ε, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτός Γενικής Διεύθυνσης ΔΕΦΚΟ και με την, εξωτερική, ε, με την Υπηρεσία Εξωτερικών Σχέσεων. Είναι ένα πολύ σημαντικό έγγραφο, είναι ένα μικρό κομματάκι, αλλά σημαντικότατο κομματάκι της, των στρατηγικών φακέλων, τους οποίους θα εξετάσουμε τους επόμενους μήνες. Έχουμε τη γενικότερη στρατηγική που έχει παρουσιάσει η ΥΠΑΤΗ εκπρόσωπος. Έχουμε τα όσα γίνονται στη Νέα Υόρκη στα πλαίσια του ΟΗΕ έτσι ώστε αυτά να μεταφερθούν και στην Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια της εξωτερικής διάστασης της αναπτυξιακής μας πολιτικής και αυτό γίνονται στα πλαίσια ε, των προσπαθειών που κάνει και ο επίτροπο Μίμητσα για, το, για την Ευρωπαϊκή Συνένεση. Εκεί συνεργαζόμαστε και μαζί σα, και έχουμε και το πλαίσιο τη Συμφωνία του Κοτονού που έχουμε συζητήσει με ιδιαίτερη ικανοποίηση και πλην ε, τη διακοπή για το καλοκαίρι. Και βέβαια Έχουμε και τα όσα θα μας πει ο Ευρωβουλευτής κ. Νόιζερ αργότερα. Έχουμε λοιπόν αυτή τη στιγμή ε, μία λίθο πάνω στην οποία θα βασίσουμε το οικοδόμημα, όχι μόνο γιατί ε, πρέπει να ατενίσουμε το μέλλον, αλλά για να ατενίσει κανείς το μέλλον πρέπει κανείς καταρχήν να αξιολογήσει το παρελθόν. Πώς ε, αξιολογούμε τα αποτελέσματα της συμφωνίας αυτής με τα 15 χρόνια εμπειρίας που έχουμε ήδη αποκτήσει για να μην δυσκολεύσω την κατανόηση που θα ε, χρειαστεί να δείξουμε σήμερα Τετάρτη πριν μετά τις διακοπές, έχω ένα PowerPoint το οποίο ελπίζω θα μας βοηθήσει. Καταρχήν, το πρώτο στοιχείο που είναι πώς μπορούμε να συνδεθούμε με τη διαδικασία της νέας εταιρικής σχέσης, πώς μπορούμε να διδαχθούμε από το παρελθόν και το τρίτο στοιχείο είναι το ότι τους περασμένους μήνες ήρθαμε σε επαφή με πάρα πολλούς από τους ενδιαφερόμενους. Πρέπει να σας πω πως διαπιστώσαμε πως υπάρχει ιδιαίτερο ζήλος για να κάνουμε αυτή την αναδρομή στο παρελθόν, για να μοιραστούμε τις εμπειρίες που έχουμε αποκτήσει και σε κυβερνητικό και σε κοινοβουλευτικό επίπεδο, αλλά και με μη καπαό όπω όπως επίσης και με την κοινωνία των πολιτών, για να δούμε τι πέτυχε η Συμφωνία Κοτονού και τι δεν πέτυχε, πού δεν πήγε τόσο καλά, πού θα έπρεπε να βελτιωθεί στο μέλλον. Γι' αυτό η αξιολόγηση είναι για μας πολύ σημαντική. Στην επόμενη διαφάνεια ε, θα σας δείξω πώς έγινε αυτή η δημόσια διαβούλευση και να σας δείξω ποιες ήταν οι πηγές μας. Καταρχήν, δημόσια διαβούλευση. Στα τέλη του περασμένου έτους κάναμε μία δημόσια διαβούλευση και λάβαμε πάρα πολλές απαντήσεις από μεγάλο φάσμα ενδιαφερομένων και τα συμπεράσματα Αυτά μπορείτε να τα βρείτε στον ιστότοπό μας. Επίσης, εξετάσαμε ε, τις πάνω από 100 στρατηγικές αξιολογήσεις που έχουμε κάνει τα τελευταία χρόνια και τις κλαδικές και τις γεωγραφικές, οι οποίες βρίσκονταν στα αρχεία της μονάδας αξιολόγησης που έχουμε και τις χτενίσαμε για να δούμε ποια είναι τα διδάγματα που μπορούμε να αποκομίσουμε χρησιμοποίησαμε και τα όσα γνωρίζουμε στα πλαίσια των υπηρεσιών μας και στη Γενική Διεύθυνση ΤΕΦΚΟ και στην ε, Trade, όπως επίσης και στην Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και στις αντιπροσωπείες μας επιτόπου, να δούμε τι γνωρίζουμε και επίσης χρησιμοποίησαμε και μια σειρά άλλων μελετών που έχουν τα κράτη-μέλη παρουσιάσει, ο ακαδημαϊκός κόσμος, οι ε, τα διάφορα ερευνητικά κέντρα, δεξαμενές σκέψεις. Και θέλω τώρα να περάσω στις βασικές διαπιστώσεις. Συμπεράσματα λοιπόν. Έχει επιτευχθεί καλή πρόοδος ε, για τους βασικούς στόχους που είχαμε θέσει. Θα σας πω περισσότερες λεπτομέρειες αργότερα. Να σας πω καταρχήν πως πρώτος η συμφωνία αυτή ε, καταρχήν ε, έχει συνεισφέρει στην εξάλληψη της ένδυας. Όχι ότι τα έχουμε καταφέρει βεβαίως, απολύτως, αλλά από την αξιολόγηση που έγινε από τους ενδιαφερόμενους, αυτή η συμφωνία, η εταιρική σχέση βοήθησε τις χώρες εταίρους να κάνουν πρόοδο στο να ε, εξαλείψουν τη φτώχεια. Δεύτερον, βελτιωμένη ενσωμάτωση των χωρών ακές στην παγκόσμια οικονομία. Οπότε η εμπορική διάσταση αυτής της ε, συμφωνίας έχει ε, επιτρέψει να πετύχουν ικανοποιητική πρόοδο. Τρίτον, έχουν ενδυναμώσει την δυνατότητα των περιφερειακών οργανισμών να αντιμετωπίσουν ε, τη διαχείριση σειράξεων. Άρα λοιπόν οι τρεις βασικοί στόχοι που είχαμε θέσει έχουν επιτύχει όλοι σημαντική πρόοδο. Το δεύτερο στοιχείο που έχει να κάνει με τα ουσιαστικά σημεία της συμφωνίας. Εκεί θα έλεγα πως τα συμπεράσματα είναι πιο μεικτά για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις δημοκρατικές αρχές και το κράτος δικαίου. Εκεί είναι πιο αμφίσιμη η κατάσταση. Μέσω του πολιτικού διαλόγου έχουμε καταφέρει και λόγω βέβαια της ε, καλύτερης χρηματοδότησης και μεγαλύτερης χρηματοδότησης ε, των 10 προγραμμάτων πλησίων να ε, ενισχύσουμε κάποιους θεσμούς, όμως όσα έχουμε κάνει δεν επαρκούν. Οι αρχές αυτές μπορεί μεν να εμφανίζονται σε μια συμφωνία που υπογράφεται και από τις χώρες εταίρους, αλλά αυτό δεν επαρκεί έτσι ώστε να υπάρχει και η πολιτική βούληση σε επίπεδο χωρών εταίρων να σεβαστούν αυτές τις αρχές. Ο διάλογος άρθρου 8 φάνηκε ιδιαίτερα χρήσιμος, πρέπει να ενδυναμωθεί. Το άρθρο 6 και αυτό χρησιμεύσε σε μια ε, σειρά περιπτώσεων και ε, για παράδειγμα στην ακτή του Λεφαντοστού ε, και στο Φίτζι και στην Κεντρική Αφρικανική Δημοκρατία το 2003, το 8 και το 5 πέτυχε αλλά έχουμε και κάποιες περιπτώσεις όπου το άρθρο αυτό δεν επέτυχε τους στόχους στους οποίους εμείς είχαμε θέσει που ήταν να εξασφαλίσουμε πως οι χώρες εταίροι θα συμμορφώνονται και θα σέβονται τις βασικές αρχές συμφωνίας. Για το μέλλον λοιπόν το σημείο αυτό θα πρέπει να το εξετάσουμε πιο προσεκτικά. Τρίτον, το, βασικό, το τρίτο βασικό συμπέρασμα της αξιολόγησης είναι πως υπάρχει μια ξεκάθαρη ένδειξη πως προσφέρουμε κάποια συγκριτικά πλεονεκτήματα. Καταρχήν η σχέση μας αυτές με τις χώρες ΑΚΕ ε, ε, δίνεται δίνει τη σταθερότητα της μακροπρόθεσμης παρουσίας μας στην περιοχή. Κάτι το ιδιαίτερα πολύτιμο. Δεύτερον, η συστράτευση της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης θεωρείται πως είναι πολιτικά ουδέτερη. Ε, το οποίο σημαίνει πως ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζονται τα κράτη-μέλη και το πώς μας βλέπουν και το γεγονός πως οι σχέσεις μας με τις χώρες ΑΚΕ βασίζονται στο ότι είμαστε Ευρωπαϊκή Ένωση σημαίνει πως δεν θεωρείται πως έχουμε κάποια και καλυμμένα συμφέροντα. Αυτή λοιπόν η ουδετερότητα με την οποία μας αντιλαμβάνονται ε, μάλλον το ότι μας αντιλαμβάνονται ως ουδέτερη δύναμη, έχει πλέον ε, και αυτό ε, σημαίνει πως ακόμα και τα κονδύλια τα οποία έχουμε προϋπολογίσει ε, αντιμετωπίζονται ως κονδύλια στα οποία μπορούν να βασιστούν, τα οποία έχουν συνέχεια και ε, δεν έχουν πολιτικό χρωματισμό. Επίσης, κρίσιμη μάζα στην ε, ε, οικονομική βοήθεια που προσφέρουμε, γιατί η συνθήκη αυτή συνοδεύεται από ένα χαρτοφυλάκιο χρηματοδότησης, το οποίο είναι ισχυρό. Επίσης, ο τρόπος με τον οποίο αυτά τα ε, οικονομικά μέσα εφαρμόζονται στην πράξη μέσω με ενό φάσματος φάσματο ε, μηχανισμών ε, και μεσών είναι κάτι το οποίο έχει εκτιμηθεί ιδιαίτερα. Η χρηματοδότηση των έργων, η στήριξη του προπολογισμού, δανεισμός κτλ. Επίσης αναγνωρίζεται το γεγονός πως έχουμε την πολιτική και τεχνική πραγματογνωμοσύνη σε κλάδους κλειδιά που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της εταιρικής σχέσης στις χώρες εταίρους. Αυτά λοιπόν είναι τα βασικά ευρήματα. Για να πω σε κάποιες λεπτομέρειες. Έχουμε τέσσερις ε, πυλώνες σε αυτή την πολιτική. Πολιτική, οικονομική, αναπτυξιακή και την πιο ε, συστημική προσέγγιση. Πολιτικά λοιπόν πορίσματα. Είναι μεγάλο πλεονέκτημα το ότι υπάρχει πλέον πολιτικός διάλογος. Είναι πρόσφατος, αλλά η αποτίμηση θεωρεί ότι είναι σημαντικό στοιχείο. Μέσω αυτής της συμφωνίας έχουμε τη βάση για τακτικό πολιτικό διάλογο με βάση το άρθρο 8 με τις χώρες με τις οποίες έχουμε αυτή την εταιρική σχέση. Ένα διάλογο που καλύπτει πολλά θέματα και κοινέ ανησυχίες. Αυτό θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό πλεονέκτημα της Συμφωνίας Κοτονού. Δεν ε, έχει πάντα τα καλύτερα αποτελέσματα, αλλά το γεγονός ότι βασίζεται στην ε, Συμφωνία μας δίνει μια νομική βάση για τη διεξαγωγή του είναι πολύ ισχυρό στοιχείο μας επέτρεψε να προωθήσουμε καλύτερη αλληλοκατανόηση των θέσεων των μεν και των δε. Οι αδυναμίες, όπως είπα, είναι ότι δεν υπάρχει πάντα πολιτική βούληση για τα ουσιώδη σημεία για την τήρηση των ουσιωδών σημείων αυτής της συμφωνίας ακόμη και αν τα έχουν προσυπογράψει όλοι για το άρθρο 96 την αποτελεσματικότητα που καθορίζεται από την πολιτική βούληση. Το άρθρο 96 λοιπόν η εφαρμογή του δεν δίνει πάντα τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα και όσον αφορά τις διατάξεις για την ειρήνη και την ασφάλεια Επίσης θεωρούμε ότι υπάρχουν σαφείς αδυναμίες. Δεν έχει πάντα λειτουργήσει όσο καλά θα θέλαμε. Τα αναφέρατε και εσείς αυτά τα θέματα στο τμήμα που αφορά τις μελλοντικέ προοπτικές και τέλος είναι μη ικανοποιητική εφαρμογή του άρθρου 13 για την μετανάστευση. Δεν χρειάζεται να σας πω περισσότερα γι' αυτό. Όλοι το αντιμετωπίζουμε καθημερινά αλλά θα πρέπει λιγάκι να διαφοροποιήσω την ε, συνολική αυτή εκτίμηση. Ε, υπάρχουν βελτιώσεις ορισμένα σημεία για τη μη διάκριση, αλλά η επανεισδοχή δυστυχώς δεν έχει εφαρμοστεί όσο θα θέλαμε. Στο σημείο αυτό η εταιρική σχέση δεν έχει λειτουργήσει όσο θα θέλαμε. Υπάρχουν πολλοί λόγοι. Πρώτα απ' όλα οι χώρες εταίροι μας έχουν προβλήματα, αλλά και εμείς δεν έχουμε δώσει αρκετή προτεραιότητα στην εφαρμογή αυτού του άρθρου στον πολιτικό μας διάλογο με αυτές τις χώρες για πολλά χρόνια. Το θέμα αυτό πρόσφατα το ανακαλύψαμε. Ακόμη και εμείς οι ίδιοι δεν μπορούμε λοιπόν να κατηγορήσουμε μια συμφωνία 15 ετούς διάρκειας τώρα θα ήταν λιγάκι ε, μικρόψυχο, αλλά οπωσδήποτε θα πρέπει να γίνουν περισσότερα στο μέλλον γι' αυτό. Το δεύτερο μεγάλο τμήμα Εμπόριο και οικονομία. Σαφώς έχουν αυξηθεί εμπορικές ροές από και προς τις χώρες ΑΚΕ. Έχουμε συνάψει συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης. Η υπογραφή και επικύρωση ε, είναι εν εξελίξη. Αλλά η ολοκλήρωση και η υπογραφή σημαίνει ότι ωφελούνται με διάφορους τρόπους ε, οι χώρες ΑΚΕ κάτι που δεν θα συνέβαινε με βάση μόνο τους κανόνες του ΠΟΕ. Και επίσης έχει αυξηθεί ο αριθμός των χωρών ΑΚΕ που συμμετέχουν στον ε, ΠΟΕ. Από την άλλη μεριά, η αποτίμησή μας δείχνει ότι η εταιρική σχέση δεν έχει δώσει ικανοποιητικά αποτελέσματα όσον αφορά την διαφοροποίηση της οικονομίας των χωρών αυτών και τη μείωση της εξάρτησης από, βασικές, ε, από μερικά βασικά προϊόντα. Βλέπουμε τώρα για παράδειγμα ότι η μείωση των τιμών αυτών των πρώτων υλών και βασικών προϊόντων έχει επιπτώσεις στις οικονομίες των χωρών αυτών. Αλλά τα στοιχεία για τις εμπορικές ανταλλαγές, συναλλαγές καλύτερα, είναι πολύ ενδιαφέροντα, είναι πολύ ικανοποιητικά. Οι εισαγωγές μας από τις χώρες αυτές έχουν αυξηθεί από το 2,8 στο 4,5. Ε, ή μάλλον 5,4. Αυτό δείχνει λοιπόν ότι έχουν αυξηθεί οι εμπορικές ροές. Τέλος, το αναπτυξιακό τμήμα της σχέσης. Ε, η αποτίμησή μας ε, αποδεικνύει ότι έχουμε συμβάλει στην εκρίζωση της φτώχειας, ούτως της φτωχειας ουτω ωστε να υπάρχει πιο ισότιμη πρόσβαση σε, στις βασικές υπηρεσίες, αύξηση της συνειδητοποίησης για περιβαλλοντικά και κλιματικά θέματα και η προώθηση της μακροοικονομικής σταθεροποίησης. Αδυναμίες, αυτά που δεν επέτυχε αρκετά το, η Συμφωνία Κοτονού, είναι φυσικά οι σειράξει και η συνεχιζόμενη ύπαρξη ε, εστιών σειράξεων. Δεν έχουμε κάνει αρκετά για να αντιμετωπίσουμε τις βασικές αιτίες των ε, συγκρούσεων. Προσπαθούμε απλώς να απαλύνουμε τις επιπτώσεις τους. Δεν έχουμε αντιμετωπίσει τις ρίζες των σειράξεων. Πρέπει να το κάνουμε στο μέλλον. Δεύτερον, δεν είχαμε αρκετή επιρροή στην ε, δικαιότερη κατανομή του εισοδήματο και σε πολύ γενικότερες ε, πολιτικο-οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες οι δείκτες που έχουμε δεν έχουν βελτιωθεί. Τρίτον, δεν έχουμε ασχοληθεί αρκετά με την ε, ανάπτυξη αύξηση του πληθυσμού καλύτερα. Υπάρχουν ε, τρομερές δημογραφικές προκλήσεις ε, σε πολλές χώρες. Θα πρέπει στο μέλλον να μας απασχολήσει περισσότερο. Και τέρον, η σταθερότητα των αποτελεσμάτων μας. Είναι ε, κάτι που ισχύει βεβαίως και για τη συμφωνία αυτή και για άλλες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες μας. Τέλος, τα μέσα που χρησιμοποίησαμε. Εξετάσαμε τα μέσα που είχαν νομικά δεσμευτικό χαρακτήρα και θεωρήσαμε ότι ήταν ε, πολύ αποφασιστική σημασία, πολύ αποτελεσματικά. Το γεγονός ότι τα βασικά στοιχεία της συμφωνίας περιέχονται σε μια νομικά δεσμευτική συμφωνία είναι κάτι που δεν ε, είναι τόσο διαδεδομένο και βλέπουμε ότι ο σχεδιασμός και η εφαρμογή των προγραμμάτων έχει προσαρμοστεί στις ανάγκες των χωρών αυτών Άρα αυτό έχει βοηθήσει την ε, αποδοχή τους από τον πληθυσμό. Αυτά ήταν θετικά. Αδυναμίες είναι ότι ο νομικά δεσμευτικός χαρακτήρας δεν είχε τα ίδια αποτελέσματα για όλα τα μέτρα, για όλους τους τομείς πολιτικής και επίσης η αποτελεσματικότητα της διαχείρισης των προγράτων, ιδιαίτερα του προϋπολογισμού, πρέπει να μας αποσχολήσει περισσότερο. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Ο ρόλος ε, των ε, εθνικών αρχών έγκρισης των δαπανών είναι πολύ σημαντικός, ούτως ώστε να υπάρχει αποδοχή, αλλά από την άλλη μεριά δημιουργεί και προβλήματα. Για παράδειγμα, σε μια συγκεκριμένη χώρα, ναι μεν συμφωνούμε με τον Υπουργό, για παράδειγμα τον Υπουργό Παιδείας ή τον Υπουργό Γεωργίας, αλλά λόγω του συστήματος του ποιος εγκρίνει τις δαπάνες, δεν αρκεί, γιατί πολύ συχνά τις, τις δαπάνες τις ε, εγκρίνει ο Υπουργός Οικονομικών. Μπορεί λοιπόν να συμφωνήσουμε με τον αρμόδιο Υπουργό για μια συγκεκριμένη πολιτική σε ένα συγκεκριμένο τομέα, πρέπει να παρέμβει και ο Υπουργό Οικονομικών. Και αυτό συχνά δημιουργεί προβλήματα. Και αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν εσωτερικές διχογνωμίες οι οποίες επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα της πολιτικής μας. Αλλά φυσικά δεν πρέπει μαζί, τα, μαζί με τα ξερά να κάψουμε και τα χλωρά. Δεν πρέπει δηλαδή να θεωρήσουμε ότι όλα είναι αρνητικά. Πολλά μπορούμε ακόμη να κάνουμε. Και αυτό σαφής ένδειξη από αυτή την προσπάθεια μελέτης ε, της αποτελεσματικότητας της εφαρμογής. Νομίζω ότι αρκετά είπα, θέλω να αφήσω χρόνο και για τους ε, συναδέλφους από τις χώρες ΑΚΕ και φυσικά και για τα μέλη της Επιτροπής σας. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ για αυτήν την ε, αναλυτική αντιμετώπιση. Έχουμε εδώ και το Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού ΑΚΕ, είναι ο Δόκτωρ Γκόμες. Καλώς ήρθατε. Ξέρουμε ότι τα θέματα αυτά είναι πολύ σημαντικά για σας. Σήμερα το απόγευμα θα ψηφίσουμε επί της εκθέσεως Νόιζερ. Δεν ξέρω αν θέλετε να μας πείτε κάτι κύριε Γενική Γραμματέα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η γραμματεία μας ε, εκτιμά το γεγονός ότι προσκλήθηκε. Σας ευχαριστεί για την παρουσία. Θα είμαι σύντομος. Και βεβαίως έχουμε και τον επόμενο πρόεδρο της Επιτροπής των ε, Πρέσβεων και απορισμένους πρέσβεις. Ευχαριστώ πολύ την Επιτροπή σας για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε αυτό το θέμα και για τη στενή συνεργασία. Θεωρούμε ότι αυτή η διαδικασία πρέπει να εμβαθυνθεί, να υπάρχει πιο στενή συνεργασία μαζί μας. Και εμείς θα έχουμε πιο στενή συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Η πρόσφατη συνάντηση κορυφής μα στο Port Moresby ήταν πολύ σημαντική. Όπως ξέρετε υπάρχει μια ομάδα επιφανών ε, προσώπων και ο, ο κύριος Ομπασάντζο θα παρουσιάσει την έκθεση σε μια ειδική εκδήλωση της ε, έκτακτη συνάντηση κορυφής Αφρικανικής Ένωση στον Τόγκο τον Οκτώβριο. Θα γίνει μια ευρύτερη λοιπόν συζήτηση για όλες τις ε, περιοχές μας και για τον ειρηνικό θα ακούσουμε λοιπόν την άποψη της ομάδας επιφανών προσώπων και είχαμε και μία ομάδα εργασίας για τις προοπτικές. Τρίτον, για την Καραϊβική θα συνεδριάσει σε επίπεδο Συμβουλίου τον Οκτώβριο το Κάρι Φόρουμ. Βλέπουμε λοιπόν ότι η διαδικασία αυτή είναι πολύ ευρεία, συμμετέχουν όλο και περισσότεροι εμπλεκόμενοι φορείς, όχι μόνο σε πολιτικό επίπεδο, ιδιωτικοί φορείς, ε, κοινωνία των πολιτών. Και επίσης, όλη μας η εργασία, όλη μας, όλες μας οι διαβουλεύσεις επιβεβαιώνουν την εκτίμηση ότι έχουμε ισχυρά θεμέλια με αυτά αποτελέσματα. Αλλά υπάρχουν και αδυναμίες, πρέπει να αντιμετωπιστούν. Αλλά και πλεονεκτήματα που πρέπει να ε, ενδυναμωθούν. Για παράδειγμα, είχαμε στον Αερόμπι την διάσκεψη UNCTAD, όπου και εμείς και η Ευρωπαϊκή Ένωση τόνισαν τη σημασία του εμπορίου και των επενδύσεων και ασχοληθήκαμε και με νέους τομείς. Πρέπει να ε, εντάξουμε και την ε, γαλάζια οικονομία που συνδέεται με την αλληλεία και την οικονομία των ωκεανών. Νέοι τομείς λοιπόν. Θα ασχοληθούμε και με αυτούς. Ε, είναι ενθαρρυντικό αυτό. Θέλουμε να εδραιώσουμε αυτά που έχουμε αλλά πρέπει να είμαστε και ιδιαίτερα επικριτικοί έναντι των αδυναμιών μας. Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις μεταξύ των χωρών, αλλά υπάρχει και αναβάθμιση κάποιων χωρών. Για παράδειγμα, από λιγότερο αναπτυγμένε χώρες, ορισμένες, όπως η δική μου η Γκάνα, είναι αναπτυσσόμενες. Δεν πρέπει να υπάρχουν ε, όμως ε, γι' αυτό το λόγο μέτρα τα οποία θα έχουν αρνητικέ επιπτώσει. Δεν είναι δυνατόν να αφαιρέσουμε κάθε είδο βοήθεια κάθε είδο επιδότηση, γιατί αυτό τραβάει το χαλί κάτω από τα πόδια μα. Θεωρούμε λοιπόν, θεωρούμε λοιπόν ότι το Αναπτυξιακό Ταμείο επίσης μπορεί να βοηθήσει. Μας βοηθάει πάρα πολύ και θέλουμε οπωσδήποτε να εκτιμήσουμε, να υπάρχει μια σωστή αποτίμηση και του τρόπου με τον οποίο λειτουργούν οι θεσμοί μας. Για παράδειγμα, οι κοινοβουλευτικοί μας θεσμοί πρέπει να βοηθήσουν, ούτως ώστε οι αποφάσεις που λαμβάνουν που λαμβάνουν από κοινού στην κοινή κοινοβουλευτική συνέλευση, στην ισο, ισομερή κοινοβουλευτική συνέλευση, πρέπει να εφαρμόζονται αποτελεσματικά. Πρόεδρος, σας ευχαριστώ και προσβλέπουμε στην περαιτέρω συμμετοχή σας όπως θα προχωρούν οι συζητήσεις. Ο Νόρμπερτ Νόιζερ που είναι ο εισηγητή μα για αυτή την πρώτη τη συμφωνία, Κοντονού. Ευχαριστώ πολύ ο κύριο Νόιζερ Λίντα. Θέλω να καλωσορίσω και πρώην μέλη της Επιτροπής μας ε, ε, που βοήθησαν εδώ και 20 χρόνια για να συναυθεί η Συμφωνία Κοτονού και τώρα ενδιαφέρονται πολύ για την αποτίμηση της ε, μέχρι τώρα πρόοδου και της περαιτέρω εξελίξης. Αγαπητέ κύριε Κούντουνς, είναι πολύ καλή αυτή η αποτίμηση των όσων επιτύχαμε μέχρι τώρα στα πλαίσια της Συμφωνίας Κοτονού για μας στο Κοινοβούλιο θα ήταν καλύτερα αυτή η αποτίμηση να είχε εκπονηθεί νωρίτερα, πριν από ένα χρόνο δηλαδή. Αλλά συνεργαζόμεθα στενά με την Κομισιόν και τώρα βλέπουμε λοιπόν μια κανονική έκθεση η οποία τονίζει και ποιες είναι οι προοπτικές συνεργασίες μεταξύ των Χρονάκια και της Ένωσης και πέρα από το 2020. Είναι σαφές από την ε, παρουσίαση ποια είναι τα θετικά και το οποίο τονίζουμε και πρέπει να τα τονίζουμε όταν καλούμε πάντα να τηρούνται οι βασικές δημοκρατικές αρχές, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου, δημιουργούμε ένα πλαίσιο Έχουμε δηλαδή μέσω της συμφωνία Κοτονού αυτό το πλαίσιο για να ζητήσουμε από τις χώρες να εφαρμόσουν αυτές τις αρχές και να καταδείξουμε και τις ευθύνες των κρατών. Πρέπει να ενισχύσουμε λοιπόν τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Γιατί αυτό έχει πολύ θετικά αποτελέσματα. Βεβαίως ε, υπάρχουν ελλείψεις ε, σε κάποιες χώρες αλλά θεωρούμε ότι αυτή η συμφωνία δημιουργεί δυνατότητες για να αντιμετωπιστούν αυτές οι ελλείψεις. Επιτύχαμε τη δημιουργία πολλών περιφερειακών μηχανισμών για να αντιμετωπιστούν οι σειράξεις. Θα μπορούσαμε να τα έχουμε πάει καλύτερα βέβαια, αλλά στην Αφρική ιδίω έχουν γίνει πολλά για την ειρήνη και την ασφάλεια με βάση την δραστηριότητα αυτών των περιφερειακών μηχανισμών, μηχανισμών αντιμετώπισης των σειράξεων. Η Συμφωνία Κοτονού βοήθησε να ενταχθούν οι χώρες αυτές στην παγκόσμια οικονομία και να βελτιωθούν οι δυνατότητες εμπορικής ε, πολιτικής και εμπορίου των χωρών αυτών. Νομίζω ότι δόθηκε πολύ οικονομική βοήθεια, στηρίξαμε προγράμματα. Αυτός ο γενικός προϋπολογισμός βοήθησε ε, να ε, βελτιωθεί η γενικότερη οικονομική κατάσταση. Μερικές βασικές υπηρεσίες, υγεία, εκπαίδευση, βελτιώθηκαν. Και αυτό πρέπει να το τονίσουμε. Υπάρχουν βέβαια δυναμίες και τις αναφέρουμε και στην εκθεσή μας και θέλουμε να αντιμετωπιστούν. Για μένα το βασικό είναι η συνεργασία μεταξύ των ε, χωρών της Ένωσης και των 79 χωρών εταίρων μας. Εκεί θα έπρεπε να μπορούμε να συνεργαστούμε όμως περισσότερο. Για παράδειγμα, αν όλοι αυτοί οι 27, 28 και 79 είχαν ενιαία θέση για παράδειγμα για τις κλιματικές διαπραγματεύσεις, θα είχαμε πλειοψηφία. Επίσης πρέπει να βελτιώσουμε την κατάσταση στον τομέα της ισότητας των φύλων. Νομίζω ότι υπάρχουν επιτεύγματα στις ε, χώρες αυτές, αλλά είναι ανεπαρκή. Και περισσότερη βιωσιμότητα χρειάζεται. Δηλαδή, οι εθνικές αρχές της χώρας αυτές πρέπει να εμένουν στην εφαρμογή των αποφάσεων. Για τον πολιτικό διάλογο, την οικονομική, εμπορική πολιτική και την αναπτυξιακή πολιτική, θέλω να τονίσω ότι δεν έχουμε αξιοποιήσει αρκετά το άρθρο 8 στην ισομερή κοινοβουλευτική συνέλευση θα μπορούσαμε να, να έχουμε επιμείνει περισσότερο σε αυτό και να καταδείξουμε τις αδυναμίες της εφαρμογής του στον τομέα ειρήνη και ασφάλεια. Δεν νομίζω ότι ανταποκριθήκαμε στις προσδοκίες. Υπάρχουν βελτιώσεις, αλλά υπάρχουν και ελλείψεις. Ιδιαίτερα σε αυτό που αναφέρθηκε για το άρθρο 13, <clears throat> που αφορά τις προκλήσεις λόγω της μετανάστευσης. Στον τομέα της εμπορικής και οικονομικής πολιτικής νομίζω ότι βοηθήσαμε την καλύτερη πρόσβαση και ένταξη των χωρών αυτών στον ΠΟΕ και η περιφερειακή συνεργασία <clears throat> σε ορισμένες περιοχές της Αφρικής οδήγησε σε περισσότερη ανάπτυξη. Αναπτυξιακή συνεργασία τώρα. Για την καταπολέμηση της φτώχειας. Επιτύχαμε πολλά μέσω αυτής της συνεργασίας. Ιδιαίτερα στον τομέα της εκπαίδευσης και της υγείας. Αλλά για την πρόληψη των συγκρούσεων πρέπει να γίνουν περισσότερα πιστεύω. Επίσης θα είμαι επικριτικός για το γεγονός ότι ότι τα κράτη-μέλη δεν συνεργάζονται παρκώς, δεν βοηθούν να υπάρχει ενωσιακή στρατηγική. Και το αναφέρει αυτό η έκθεση και το διαπίστωσα και εγώ. Πολλοί λένε θέλουμε περισσότερο να έχουμε μια αυτόνομη πολιτική δική μας. Αλλά θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε ότι μέσω αυτού του κοινού νομοθετικού πλαισίου μπορούμε να κάνουμε περισσότερο. Θα έπρεπε να το αξιοποιήσουμε περισσότερο μέσω περισσότερης περιφερειακής συνεργασίας. Κάτι άλλο επίσης, που είναι βασικό για όλα τα όσα προανέφερα. Είναι το θέμα της συμπεριφοράς της ε, Κίνας και των Ηνωμένων Πολιτειών εάν είχαν μια τέτοια οικονομική συμφωνία όπως Κοτονού. Θα έγκλειφαν τα δάχτυλά τους ε, αν είχαν τη δυνατότητα μια τέτοια συμφωνίας. Πρέπει να είναι σαφές τι πλεονέκτημα λοιπόν έχουμε και πόσο σημαντικό είναι να συνεχίσουμε να έχουμε ένα τέτοιο πλεονέκτημα, μια τέτοια συμφωνία και μετά το 2020. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Τρεις ε, συνάδελφοι έχουν ζητήσει μέχρι τώρα το λόγο. Χαουτάλα, Λίντς και Γκέπελς. Ε, α, και η Λόλα, όχι δεν θέλω να μιλήσει. Η κυρία Μαρία Χόιμπερ. Ευχαριστώ, Λίντα. Ευχαριστώ, κύριε Ντούνς. Το ερώτημα ήταν πόσο σημαντική ήταν και είναι αυτή η συμφωνία. Είναι καλή βάση για τη συνεργασία. Είναι ένα καλό πλαίσιο για να βοηθήσουμε αυτές τις χώρες να έρθουμε σε επαφή μαζί τους για να υπάρξει αναπτυξιακή συνεργασία. Και τι είναι καλή αναπτυξιακή συνεργασία. Θεωρώ ότι από τους τρεις πυλώνες, πολιτικός διάλογος, εμπόριο και αναπτυξιακή συνεργασία, η αναπτυξιακή συνεργασία έχει λειτουργήσει σωστά. Για τους άλλους δύο πυλώνες ε, έχω περισσότερες αμφιβολίες. Ε, τα αναφέρατε κι εσείς. Ο πολιτικός διάλογος είναι πολύ πρόσφατος. Και εσείς ε, είπατε ότι δεν λειτουργήσε πάντα πολύ καλά. Παρ' όλα αυτά βοήθησε την ε, αλληλοκατανόηση. Συμφωνώ. Για το εμπόριο. Ελπίζω να σας κατάλαβα καλά. Είπατε ότι η αύξηση αυτή του εμπορίου ήταν από εκείνους προς εμάς. Όχι προς την άλλη κατεύθυνση και προς τις δύο κατευθύνσεις. Αυτή είναι η ερώτησή μου. Αυτή η αύξηση των ε, συναλλαγών είναι κυρίως εξαγωγές των χωρών και προς εμάς ή πάει και προς την άλλη κατεύθυνση. Γιατί η εμπορική συμφωνία επιτρέπει και τις δύο κατευθύνσεις. Έχουν ανοίξει οι χώρες αυτές τις αγορές τους προς εμάς. Αλλά έχουν τόσες δυσχέρειες. Και βλέπουμε ότι η διαφοροποίηση της οικονομίας τους δεν έχει επιτύχει επαρκώς. Οι χώρες αυτές εξακολουθούν να είναι αδύναμες γι' αυτό το λόγο και η ευημερία τους δεν έχει βοηθηθεί. Αυτό θεωρώ ότι είναι μεγάλο πρόβλημα. Γιατί είναι προς το κοινό μας συμφέρον να ωφεληθεί ο πληθυσμός των χωρών αυτών από αυτή τη συμφωνία. Και δεν θεωρώ ότι έχει επιτευχθεί επαρκώς. Πρέπει πολλά να κάνουμε ακόμη για αυτό το θέμα. Ιδίως στην Αφρική. έχει ξεκινήσει η διαδικασία ευρω, ε, συγγνώμη, αφρικανικής ενοποίησης, της δημιουργίας μιας ε, εσωτερικής αγοράς, πρέπει να προσέξουμε να μην την παρεμποδίσουμε μέσω των δικών μας εμπορικών συμφωνιών, να τους δώσουμε τη δυνατότητα να προστατεύσουν κάπως ε, τις αγορές τους, κάποιου προστατευτισμού. Με επ' αυτού λοιπόν είμαι κάπως επικριτική. Άλλη ερώτηση. Κάνατε μια αποτίμηση του παρελθόντος και του πώς είναι τώρα η κατάσταση, αλλά δεν μας είπατε αρκετά για τις προοπτικές. Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Διαχείρισης ε, Αναπτυξιακής Πολιτικής εξεπώνησε μια έκθεση με τέσσερα σενάρια. Ποιο από αυτά ε, προτιμάτε εσείς και η γενική σας διεύθυνση. Πώς δηλαδή πρέπει να προχωρήσουμε. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με βάση αυτό το παλιό πλαίσιο ή θα κάνουμε πιο συγκεκριμένη δουλειά, θα διαφοροποιήσουμε ανάλογα με τις περιφέρειες ή ακόμη και με τις ε, μεμονωμένες χώρες ή και με τους κλάδους πολιτικής με τους οποίους ασχολούμεθα. Παρακαλώ, μπορείτε να μας πείτε λίγο περισσότερα για την ε, μελλοντική σας πολιτική πώς τη βλέπετε. Και ακόμη, το Νοέμβριο θα υπάρξει μια ανακοίνωση της Κομισιόν, από ό,τι κατάλαβα. Θα θέλουμε να μας πείτε και πώς συνδυάζεται με την προοπτική του Brexit. Γιατί το Ηνωμένο Βασίλειο είναι από τους σημαντικούς, σημαντικούς χρηματοδότες του Κοτονού. Τι θα γίνει με αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντική αυτή η συζήτηση γιατί ε, η αξιολόγηση που κάνουμε καθώς επίσης και ο τρόπος με τον οποίο αποτιμούμε τα 16 χρόνια ε, της Συμφωνίας Κοτονού είναι θέματα πολύ σημαντικά και προς τα έξω αλλά κυρίως για μας εδώ στο εσωτερικό μας γιατί και στο παρελθόν ε, έχουμε διαπιστώσει αποκλήσεις ερμηνείας ορισμένων αποτιμήσεων κυρίως από πλευρά ε, του ελεγκτικού συνεδρίου. Έρχονται λοιπόν οι εκπρόσωποι του ελεγκτικού συνεδρίου και εν τέλει διαπιστώνουμε ότι η δικιά μας ερμηνεία ήταν η σωστή και ε, επομένως αυτή θα ήταν η καλύτερη ερμηνεία απέναντι σε άλλες ε, ε, διαφορετικές οι οποίες όμως κυριαρχούν στον τύπο. Νομίζω λοιπόν ότι είναι πολύ σημαντικό εδώ στην Επιτροπή μας αλλά και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να έχουμε κοινή αποτίμηση έτσι ώστε να έχουμε μια καλή εναρκτήρια θέση σε σχέση με, την, με αυτό που θα ακουστεί προς τα έξω. Δεύτερο, όταν περάσαμε από τη Λομέ στην ε, Συμφωνία Κοτονού είχαμε υποσχεθεί στους εαυτούς μας ότι θα κάνουμε πολλαπλές ε, ε, πρόοδους ή βελτιώσεις, βελτιώσεις των προγραμμάτων ε, δηλαδή θέλαμε να συμπεριληφθούν νέοι ε, εκπρόσωποι, κυρίως κοινωνίας των πολιτών και του ε, ιδιωτικού τομέα, ανάπτυξη των επιδόσεων, να έχουμε μία ειδική προσέγγιση αναχώρα, καθώς επίσης και μία αποκεντρωμένη διοίκηση και διαχείριση. Νομίζω ότι στα περισσότερα από αυτά τα σημεία έχουμε μάλλον επιτύχει, έστω και αν πολλές φορές ε, οι ε, επιτυχίες μας ε, πρέπει ακόμα να επιβεβαιωθούν κυρίως απέναντι σε νέους πρωταγωνιστές και βεβαίως εάν αν δούμε και αν συνυπολογίσουμε πόσο μεγάλα ήταν τα εμπόδια τα οποία η πλευρά και είχε θέσει για την συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στην αρχή και αν λάβουμε υπόψη μας το γεγονός ότι πλέον η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών είναι εκ των μπορούμε να πούμε ότι έχουμε κάνει σημαντικές προόδους αλλά βεβαίως ακόμα πολλά πρέπει να γίνουν όσον αφορά Ε, τα, τα μεγάλα πολιτικά διακυβεύματα, οικονομικά ε, ε, και βεβαίως ακόμα υπολείπεται η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών. Όσον αφορά την τυποποιημένη προσέγγιση, είναι γεγονός ότι πλέον έχουμε προσέγγιση ιδιαίτερη αναχώρα. Αυτό είναι πολύ καλό. Ε, τώρα εγώ θα ήθελα να ασχοληθώ περισσότερο με τα αρνητικά στοιχεία, τα οποία, η σημεία τα οποία ανέφερε ο κύριος Κούνς ο κύριος Ντόνουσε, συγγνώμη. Νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, ε, γιατί δεν ασχοληθήκαμε αρκετά με την ε, δημογραφική αύξηση ε, νομίζω λοιπόν ότι εδώ θα πρέπει να δούμε βέβαια το θέμα και από τις δύο πλευρές ξέρουμε ότι ε, είναι πολύ ευαίσθητο θέμα και δύσκολο να το συζητήσουμε με την, ε, με την άλλη πλευρά και ακόμα και στη δικιά μας Επιτροπή πολύ λίγο προχωράμε όταν ξεκινάμε συζήτηση για οικογενειακό προγραμματισμό ακόμα και όταν μιλάμε και για την δημόσια υγεία, την, τους ε, με, ε, ε, υπό την επιτήρηση γιατρού λοιπά Επομένως είναι πάρα πολύ προσεκτικές και διστακτικές οι χώρες αυτές να συζητήσουν για τα θέματα αυτά. Ε, όσον αφορά όμως ε, το διεθνές δίκαιο, νομίζω ότι έχουμε προχωρήσει και όλες αυτές οι δίκες ε, στο δικαστήριο της Χάγης ακριβώς αυτή την πρόοδο καταδεικνύουν. νομίζω ότι είναι καλό να δούμε ότι έχουμε κάνει πολλά βήματα στα πλαίσια των χωρών και έχουμε κάνει πολλά βήματα όσον αφορά και προόδους. Βεβαίως μπορούμε να προχωρήσουμε ακόμα περισσότερο και έχουμε προχωρήσει περισσότερο με ορισμένε χώρε ΑΚΕ παρά με ε, τι Ηνωμένε Πολιτείε ή άλλου ε, ε, παραδοσιακού συμμάχου μα. Τώρα, όσον αφορά την φτώχεια, εδώ υπάρχει ένα πραγματικό πρόβλημα. Η διεθνή κοινότητα θέλει να δώσει λύση στα πλαίσια κυρίω των στόχων τη βιώσιμη ανάπτυξη. Νομίζω ότι δεν έχουμε λόγο και δεν έχουμε έχουμε ε, καμία δικαιολογία να μην κάνουμε ε, κάτι γι' αυτό και να βοηθήσουμε και τους εταίρους στην Αφρική. Αλλά υπάρχει και ένα άλλο πρόβλημα το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Το δημόσιο χρέος των χωρών ήταν ε, πραγματικά μεγάλο πρόβλημα στη δεκαετία του 2000. Το πρόβλημα αυτό σε πολύ μεγάλο βαθμό έχει μειωθεί, αλλά τώρα ξανα, ξαναπαίρνει ανησυχητικές διαστάσεις. Αυτό δεν ε, ε, μεταφέρεται καλά νομίζω στις ε, αξιολογήσεις γιατί ενώ έγιναν καλές, καλά βήματα τελικά ξανά έχουμε πρόβλημα. Εδώ ένα άλλο σημείο στο οποίο θα ήθελα να ε, αναφερθώ είναι ε, αυτό το θέμα της διεθνούς συνεργασίας, της μεγάλες διασκέψεις, όπου διαπιστώνω ότι δεν υπάρχει ενιαία θέση ανάμεσα στις χώρες ε, και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει μια έλλειψη συνεργασίας και αλληλεγγύης στις μεγάλες διασκέψεις. Και πρέπει να πω ότι στην τελευταία διάσκεψη ε, τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, τα λόγια της Κομισιόν και τα λόγια των εκπροσώπων ε, των των χωρών ΑΚΕ είχαν ε, και αναφέρθηκαν σε κοινέ στρατηγικές, σε κοινού ε, προσανατολισμούς. Νομίζω ότι οι μεγάλες διαφορές ε, υπάρχουν ανάμεσα στις πιο αναπτυγμένες χώρες ΑΚΕ και στις λιγότερο. Νομίζω ότι αυτή είναι μια διαπίστωση την οποία είχαμε κάνει και στην Τόχα και η οποία είναι ιδιαίτερος λυπηρή συμφωνώ μαζί σας ε, ότι ε, στην ουσία το πρόβλημα είναι ότι δεν ασχοληθήκαμε αρκετά και δεν αντιμετωπίσαμε αρκετά τις ε, ε, ιδιαιτερότητες των αφρικανικών χωρών. Πάντως, σε γενικές γραμμές μπορώ να πω ότι έχουμε κάνει πολλά καλά πράγματα, είχαμε καλά αποτελέσματα, βεβαίως μπορούμε να κάνουμε περισσότερα και βεβαίως θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με το Brexit, με ποιο τρόπο αυτό μπορεί να επηρεάσει την Συμφωνία Κοτονού και βεβαίως να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε και να σκεφτόμαστε τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να συνεργαστούμε. Ε, ευχαριστώ πολύ. Ο συνάδελφο ευχαριστώ ε, πολύ ε, για τα στοιχεία τα οποία μας δώσατε όσον αφορά την αξιολόγηση, αλλά ευχαριστώ και τους συναδέλφους οι οποίοι αναφέρθηκαν σε πολύ σημαντικά θέματα. Εγώ θα ήθελα να αναφερθώ σε κάτι ειδικό το οποίο αναφέρατε στην παρουσίασή σας. Ε, δηλαδή διαπιστώσατε κάποιες, κάποιες δυσκολίες όσον αφορά την εφαρμογή των νομοθετικά δεσμευτικών διατάξεων και ότι δεν υπάρχει ίδια και σωστή εφαρμογή εφαρμογή παντού. Μπορείτε να μας πείτε λίγο ε, περισσότερα ε, γι' αυτό, τι σημαίνει ε, όσον αφορά τα υφιστάμενα θέματα, οι υφιστάμενες διαστάσεις, αλλά και για καινούργια θέματα, όπως ας πούμε αυτό της υφαντουργίας. Επίσης, το θέμα της χρηματοδότησης της ανάπτυξης ε, ε, ίσως θα μπορούσε να ενταχθεί το θέμα αυτό ε, στην συνολικότερη διαδικασία κοτονού, δηλαδή να δούμε πώς η αναπτυξιακή βοήθεια ε, και πώς τα αναπτυξιακά προγράμματα μπορούν να προωθηθούν καλύτερα. Ας πούμε, όσον αφορά την ε, κλιματική αλλαγή και το Ταμείο για το Κλίμα, ε, ίσως θα μπορούσε να γίνει πιο διευρυμένη αυτή η διαδικασία. επίσης, Ε, επίσης, αν κατάλαβα καλά, λέτε ότι θα υπάρξουν κάποιες ε, περικοπές όσον αφορά ε, το εμπόριο ή κάποια μείωση. Επίσης, κάποια συγκεκριμένα στοιχεία όσον αφορά το εμπόριο, όσον αφορά το κλίμα. Εγώ ήμουνα στην διάσκεψη της και συζητήθηκε το θέμα αυτό. Δηλαδή, πώς μπορούμε να διευθετήσουμε τα θέματα αυτά έτσι ώστε να προχωρήσουμε όσον αφορά την διάσκεψη των ε, Ηνωμένων Εθνών ε, για τις κατευθυντήριες αρχές για την ανάπτυξη και πώς μπορούμε να εντάξουμε τα θέματα αυτά στην ε, συνολική διαδικασία αλλά και το να δούμε τι, τι έρχεται και μετά, τι θα ακολουθήσει μήπως θα μπορούσαμε να ξανασκεφτούμε με διαφορετικό τρόπο όλες τις ε, αρχές, ε, να δουλέψουμε όλοι μαζί έτσι ώστε να μπορέσουμε να επιτύχουμε ε, τους στόχους, έτσι ώστε αυτοί οι στόχοι να μην είναι έτσι λίγο εθεροβάμονες ή να μην είναι πολύ υψηλοί οι στόχοι, αλλά να γίνουν στόχοι πραγματικοί και απτοί. Νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και ίσως θα πρέπει να δούμε με ποιο τρόπο θα μπορέσουμε να ενισχύσουμε την ε, ικανότητά μας, ε, το δυναμικό μας, έτσι ώστε να ε, προωθηθούν όλα αυτά και να μπορούμε και να τα ελέγχουμε. Ευχαριστώ πολύ. Χάιντι Χαουτάλα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Έχω την εντύπωση ότι η παρουσία των χωρών και σε αυτήν την συνεδρίαση είναι πάρα πολύ σημαντική έτσι ώστε να καταλάβουμε ε, και την δική τους άποψη. Εγώ ε, θεωρώ ότι γενικά έχουμε βεβαίως μια ε, γενική γραμμή θετική αξιολόγηση έστω και αν εξακολουθούν να υπάρχουν κάποια αρνητικά στοιχεία τα οποία και οι ίδιες χώρες ΑΚΕ και ο πρόσωπο της Κομισιόν και οι συνάδελφοι έχουν αναφέρει. Πιστεύω ότι θα πρέπει να διατηρήσουμε αυτά τα θετικά στοιχεία της ε, ε, Συμφωνίας ε, Κοτονού, εντάσσοντας αυτήν και νέες ιδέες και νέες πρακτικές. Η περιφερειοποίηση νομίζω ότι είναι η λέξη κλειδί και ο τρόπος με τον οποίο θα πρέπει προχωρήσουμε παρόλα αυτά. Θεωρώ ότι θα πρέπει η συνεργασία μας και με την Καριφόρο και με την Αφρική, με τις χώρες ΑΚΕ θα πρέπει να παρέχει και ένα γενικότερο πλαίσιο όμως. Το Κοινοβούλιο έχει ιδιαίτερο υπογραμμίσει την ανάγκη ενδυνάμωσης του πολιτικού διαλόγου. Εν τέλει θεωρώ ότι πολλά προβλήματα μπορούν ε, να λυθούν με μεγαλύτερη διαφάνεια, με μεγαλύτερο απολογισμό ε, και μεγαλύτερη σαφήνεια να πω ότι έχουμε και κάποιες ε, τροπολογίες στην έκθεση, κυρίως από την Λόλα Σάντσες Καλεντέη. Και αυτά τα πολιτικά ζητήματα θα πρέπει να υπογραμμιστούν. Ε, γνωρίζουμε ότι η Αφρική έχει κερδίσει ε, ε, από την ένταξη των γυναικών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Αναφέρθηκε επίσης ότι η Συμφωνία Κοτονού δεν είχε ικανοποιητικά, πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα ε, στις ε, κοινέ θέσει ε, στη, επί διεθνών θεμάτων και στα διεθνή φόρα. Πιστεύω λοιπόν ότι σε αυτό το σημείο πολλά μπορούν ακόμα να γίνουν. Έχω την αίσθηση ότι αυτά τα φόρα τα οποία έχει, προσθέσει ή έχει προσφέρει η Συμφωνία Κοτονού δεν έχουν χρησιμοποιηθεί αρκετά έτσι ώστε αυτές οι 79 χώρες ΑΚΕ και οι 28 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να έχουν μια κοινή θέση όσον αφορά ε, θέματα όπως είναι η κλιματική αλλαγή, όπως είναι η μείωση της ε, ένδυας. Ε, η κοινοβουλευτική συνέλευση είναι πολύ σημαντική. Εγώ μάλιστα είμαι και αντιπρόεδρος της Euronest που βεβαίως είναι μια διαφορετική συνέλευση, αλλά παρόλα αυτά πρέπει να πω ότι αυτού του είδους οι κοινοβουλευτικές συνελεύσεις θα πρέπει να μεταρρυθμιστούν γιατί δεν είναι αρκετά ελκυστικές πλέον. Ε, κυρίως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις πολύ λίγο ενδιαφέρον έχουν δείξει για να είναι παρούσες ε, στις διαδικασίες μας. Επομένως θα πρέπει να υπάρξει ε, μεταρρύθμιση ε, και νομίζω ότι όλοι μπορούμε να μάθουμε ο ένας από τον άλλον εμείς που συμμετέχουμε σε τέτοιου είδους πολυμερείς σχηματισμούς. Ε, επίσης ε, θα πρέπει να ε, δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε εμείς να στηρίξουμε μεταρρυθμίσεις του δικαστικού τομέα, της ισότητας των φύλων και τα λοιπά στις χώρες με τις οποίες έχουμε επαφή. Θα πρέπει οπωσδήποτε αυτού του είδους οι κοινοβουλευτικές συνελεύσεις να γίνουν πιο ζωντανές. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Σφέν, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Ντόνς ε, για την ε, παρουσίασή του, αλλά και τους ε, συναδέλφους για τα όσα είπαν. Είναι πολύ σημαντικό να δούμε ποια είναι τα ισχυρά και ποια είναι τα ασθενή στοιχεία της ε, συνεργασίας μας με τις χώρες αυτές. Ε, και ο συνάδελφος Νόρμπερτ επίσης πολλά σωστά είπε όσον αφορά την ενίσχυση της ε, συνεργασίας και όσον αφορά τις προοπτικές εργασίες και συνεργασίες με τις χώρες αυτές. Τώρα, όσον αφορά την διαδικασία post είναι σημαντικό να δούμε ποια είναι τα στοιχεία επί των οποίων θα πρέπει ε, να εστιάσουμε την ε, προσοχή μας ε, γιατί επί του οποίου, και το έγγραφο επί του οποίου θα εργαστεί ο Νόρμπερτ. Το θέμα της διασύνδεσης και των διασυνδέσεων γενικά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρόεδρος, να κάνω και εγώ ορισμένα σχόλια. Εσείς καταδείξατε κάποια από τα σημαντικά στοιχεία τα οποία θα πρέπει ε, να ληφθούν υπόψη. Θέματα ασφάλειας τα οποία είναι πάντα επίκαιρα. Αναρωτιέμαι όμως εάν ο τρόπος με τον οποίο ε, ε, αναφερόμαστε στην ασφάλεια ε, πριν, στα πλαίσια της Κοτονού μετά πριν από ορισμένα χρόνια και όταν αναφερόμαστε σε λύση συγκρούσεων κτλ. Αναρωτιέμαι αν έχουν την ίδια διάσταση τώρα γιατί εδώ έχουν προσθεθεί νέα στοιχεία και επομένως με διαφορετικό τρόπο πλέον πρέπει να βλέπουμε τα θέματα της ασφάλειας και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν αυτά να αντιμετωπιστούν στα πλαίσια των εταιρικών σχέσεων. Το θέμα της δημογραφικής αύξησης επίσης είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Οι αριθμοί, ιδιαίτερα στην ε, ε, Αφρική, ε, είναι πάρα πολύ μεγάλοι. Ξέρουμε ότι τι έγινε και το 19ο αιώνα στην στην Ευρώπη πώς αντιμετωπίστηκε το θέμα της αύξησης του πληθυσμού με την ε, μετανάστευση. Ε, γνωρίζουμε ε, πώς αντιμετωπίστηκε η φτώχεια και τους προηγούμενους Αιώνε. Ε, ε, βεβαίως δεν μπορεί να απαντηθεί απλά αυτό το περίπλοκο ερώτημα, αλλά παρόλα αυτά δεν θα πρέπει να το αφήσουμε ε, στην άκρη ή να το παραμελήσουμε όπω κάναμε μέχρι τώρα. Πολλέ αναλύσει έχουν γίνει ε, που αναφέρονται σε πολλέ λύσει, αλλά νομίζω ότι ο διάλογο είναι το πιο σημαντικό. Γι' αυτό άλλωστε θα έχουμε και μια κοινή συνεδρίαση με την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων που ακριβώ θα έχει θέμα την μετανάστευση. Νομίζω ότι αυτή είναι μία ε, προτεραιότητα γιατί πρόκειται για φαινόμενα τα οποία γνωρίζουμε εμείς ε, ε, πολύ καλά οι Ευρωπαίοι. Άλλο θέμα. Μία από τις επικρίσεις ε, που αφορούν ε, την ε, Κοτονού και τον τρόπο χρηματοδότησης είναι η έλλειψη ευελιξίας. Μιλάμε για τα προγράμματα τα οποία αφορούν συγκεκριμένες χώρες, αλλά όταν παρουσιάζεται κάποια κρίσιμη κατάσταση, η επίκριση που αναφέρεται, που ακούγεται, είναι ότι δεν έχετε τη δυνατότητα να αντιδράσετε άμεσα. Πρόκειται για ένα θέμα το οποίο επανέρχεται, ίσως θα πρέπει να ε, υπάρξει μεγαλύτερη ε, ευελιξία. Ε, τώρα όσον αφορά τις λύσεις που προτείνονται, εγώ είμαι λίγο σκεπτική γιατί ωραία μπορούμε να δημιουργούμε ταμεία, αλλά εάν δεν χρηματοδοτούνται, δεν ενισχύονται τα ταμεία αυτά, τότε δεν έχουν έννοια. Και βεβαίω εμείς έχουμε και ξεκινήσει και μια συζήτηση με τις χώρες ΑΚΕ σχετικά με χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία είναι ειδικά σχεδιασμένα σχεδιασμένα για να αντιμετωπίσουν ειδικά προβλήματα. Ε, νομίζω ότι ένα άλλο ζήτημα είναι ότι όλες οι συζητήσεις γίνονται με πολύ γραφειοκρατικό, γραφειοκρατικό τρόπο σε επίπεδο ε, κυβερνήσεων, σε επίπεδο κυβερνητικών εκπροσώπων, ε, αλλά στην ουσία δεν καταφέρουμε να συζητήσουμε αυτά τα βασικά φλέγοντα θέματα τα οποία βρίσκονται στα χείλη όλων και μπορεί να προχωρήσουμε έτσι κάνοντας κάποιες συζητήσεις μακροσκελής και που όμως ε, ε, ε, εν τέλει δεν, δεν γεννούν συγκεκριμένο αυτό αποτέλεσμα. Νομίζω ότι θα πρέπει να αλλάξουμε λίγο αυτή την πολιτική έτσι ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα πολύ σοβαρά και φλέγοντα ζητήματα. Δεν ξέρω εάν κάποιος άλλος συνάδελφος θέλει το λόγο. Ναι, ο κύριος Πρέντα. Παρακαλώ κύριε Πρέντα. Ε, σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Δυστυχώς ε, έπρεπε να είμαι σε άλλη επιτροπή και δεν άκουσα την ε, κεντρική παρέμβαση του κυρίου Ντόνς, αλλά πάντως διάβασα τη σύνοψη της παρουσίασής σας. Και θα ήθελα να σας υποβάλω ένα ερώτημα γιατί είμαι και ε, μόνιμος συζητητής του Κοινοβουλίου όσον αφορά την συνοχή των αναπτυξιακών πολιτικών. Ρωτώ λοιπόν εάν η Συμφωνία Κοτονού έχει λάβει υπόψη ε, ε, αυτήν την πολιτική για την συνοχή ε, των αναπτυξιακών πολιτικών, γιατί θεωρώ ότι μεταξύ των δύο υπάρχει μεγάλη συνάφεια και άλλωστε μόνο εάν οι στόχοι της Ατζέντα 2030 εφαρμοστούν θα μπορέσει και η πολιτική για τη συνοχή των αναπτυξιακών πολιτικών η στρατηγική αυτή να έχει έννοια. Ε, στις τροπολογίες μου λοιπόν για το μέλλον των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και μετά το 2020 αναφέρθηκα στην ε, ανάγκη να υπάρξουν συνεισηγητές της, στην Κοινοβουλευτική Ισομερή Συνέλευση. Αυτή είναι η ερώτησή μου, αν υπάρχει συσχέτιση και συγγνώμη μια ακόμα φορά που έφτασα άργο πορημένος. Ξέρω πως ο πρέσβης των Αφρικαν... Ε, της ε, Επιτροπής για την Επιτροπή της και θέλει να πάρει ε, το λόγο. Λέγομαι πρέσβης Ισμπέλ και εκπροσωπώ τέσσερα μικρά νησιά στην Ανατολική Καραϊβική αλλά έχω και την Προεδρία της Επιτροπής ε, Πρέσβεων για το συγκεκριμένο εξάμεινο. Θα ήθελα να σταθώ στην πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση που μας παρουσιάστηκε πριν από λίγη ώρα από τους συναδέλφους στην ΤΕΦΚΟ και να σας πω πως τα σχόλιά μας θα είναι στοχευμένα στις χώρες στις οποίες εγώ εκπροσωπώ. Βεβαίως ε, δεχόμαστε απερίφραστα πως όταν κανείς εξετάσει και την εταιρική σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και με τα δικά μας μέλη που βρίσκονται από αυτήν την πλευρά των νεδράνων, δεν είμαστε ε, παρόμοια κράτη ούτε ε, σε μέγεθος ούτε σε πληθυσμό ότι οι δείκτες πολλές φορές ε, δείχνουν τη διαφορά μας και δεν μπορούμε τα αποτελέσματα τα οποία πετυχαίνουμε να είναι ομοιογενή γιατί βεβαίως ως οικογένεια είμαστε ομοιογενείς. Ε, χρειάζεται αλληλεγγύη αλλά Έκανα αυτή την εισαγωγή γιατί θα ήθελα να κάνω δύο-τρία σχόλια. Καταρχήν, εμπόριο και οικονομία. Θα ακούσατε τόσο είπαν οι συνάδελφοι από την ΤΕΦΚΟ, ότι το γεγονός πως η συμφωνία αυτή αποτέλεσε ένα πολύ καλό καταλήτη για την ενισχυμένη, το ενισχυμένο εμπόριο μεταξύ της περιοχής μας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η δική μας η εμπειρία από την περιοχή της Καραϊβικής είναι μάλλον κάπως διαφορετική. Είμαστε η πρώτη ομάδα η οποία υπέγραψε μια τέτοιου είδους συμφωνία εταιρικής σχέσης και στην αναθεώρηση που έγινε πριν από 1,5 χρόνο, δηλαδή στα 5 χρόνια της ε, εφαρμογής, έδειξε πως ήταν πολύ μικρές, ε, μικρά τα βήματα που έγιναν. Τώρα, Καταλαβαίνουμε πολύ καλύτερα τους κανονισμούς, τους κανόνες, έχει οικοδομηθεί το δυναμικό που έχουμε στο χώρο, αλλά αν κοιτάξουμε τα απτά αποτελέσματα επιτόπου, θα διαπιστώσουμε πως αυτά ήταν μάλλον φτωχά και η προσδοκία μας είναι στον επόμενο γύρο να έχουμε σημειώσει πρόοδο σε κάποιες περιοχές. Οι πολύ μικρές δικές μου χώρες συμμετείχαν στις διαπραγματεύσεις που έγιναν στα πλαίσια ε, του ε, Φόρουμ για την Καραϊβική υποστηρίζοντας την εξή σκέψη. Εμείς παράγουμε υπηρεσίες, όχι εμπορεύματα και έχουμε πληθυσμούς από 185.000 μέχρι 50.000 στα μικρά νησιά μας. Αυτή είναι η δική μας πραγματικότητα και αυτό που μας ε, ενδιαφέρει ιδιαίτερα ήταν η διευκόλυνση των ταξιδιών, ε, ο πολιτιστικός κλάδος, ο κλάδος της πολιτιστικής δημιουργίας, ε, οι υπηρεσίες και να μπορούμε να ερχόμαστε στην Ευρώπη όχι για να μείνουμε, αλλά να μπορούμε να αναδείξουμε το πολιτιστικό μας πλούτο. Και εκεί δεν έγινε το παραμικρό βήμα στα πλαίσια της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης. Άρα λοιπόν εκεί τους στόχους δεν τους πετύχαμε. Τώρα μας έχουν συμβουλεύσει να διαπραγματευτούμε σε ε, εξατομικημένο επίπεδο με την Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή ανά και για τους δικούς μας δημιουργούς και καλλιτέχνες να πετύχουμε μια εξαίρεση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως ε, στέκομαι στο σημείο αυτό γιατί δυστυχώς εδώ δεν πετύχαμε ε, τα όσα ε, σε αναπτυξιακό επίπεδο στον κλάδο αυτό μας είχε υποσχεθεί αυτή η συμφωνία. Ένα άλλο σημείο το οποίο δεν συζητήσαμε σήμερα το πρωί, αλλά έχουμε δει σε άλλα βήματα, είναι η κλιμάκωση. Και όπως και πολλές χώρες ΑΚΕ, είμαστε πλέον όχι χώρες φτωχές, αλλά χώρες οι οποίες έχουν πετύχει ένα βαθμό ευημερία και κάποιου πλούτου και αυτό μέσω των δικών μας, των μας πρωτοβουλειών αλλά και στηριζόμενοι από την εταιρική σχέση μεταξύ ημών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάτι το οποίο είναι πολύ πετυχημένο, πολύ ζωντανό. Αλλά το να χρησιμοποιούμε το ΑΕΠ για πολύ μικρά κράτη νησιά που και να το χρησιμοποιούμε ως δείκτη για το κατά πόσο είμαστε τροτά ή ανθεκτικά ή όχι δεν νομίζω πως είναι ένας δείκτης αναφορά αναφορά στον οποίο θα έπρεπε να χρησιμοποιούμε. Γιατί για μας το ένιγμα είναι πώς θα τα καταφέρουμε. Δεν είμαστε αρκετά φτωχοί ώστε να μας ε, προσέξουμε τον ιδιαίτερο αυτό τρόπο, αλλά δεν είμαστε και αρκετά πλούσιοι ώστε να τα καταφέρουμε μόνοι μας. Δηλαδή, ε, τροπικοί ε, κυκλώνες για παράδειγμα που χτυπάνε τα μικρά ε, νησιά και στην περίπτωση αυτή δεν αντέχει η οικονομία μας. Την μετά την Κοτονού περιοχή θέλουμε να μπορούμε να έρθουμε σε άμεση επαφή με τους ομολόγους μας στο γραφείο του Επιτρόπου Μίμητσα για παράδειγμα για την διαπραγμάτευση νέων ε, εργαλείων που θα αντιμετωπίζουν την πραγματικότητα αυτού που είμαστε. Ούτε αρκετά πλούσιοι, ούτε αρκετά φτωχοί και βεβαίως πάντα ε, χρειαζόμαστε κάποιο είδους ε, συστηματική σχέση μαζί σας για να προοδεύσουμε. Ναι, και μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα το να ενισχύσουμε τον ιδιωτικό κλάδο, καταγράφουμε πως υπάρχουν τα ε, εργαλεία από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έτσι ώστε να ανθίσει ο κλάδος αυτός. Όμως δεν μπορούμε να έχουμε την ίδια λύση που θα εφαρμόζουμε σε όλους, τουλάχιστον στο, στα εργαλεία που χρησιμοποιούνται. Αν δείτε λοιπόν το 86% των κρατών της ε, ε, Ανατολικής Καραϊβικής, όπου οι επιχειρήσεις ε, απασχολούν από ένα μέχρι τέσσερα οικογενειακά μέλη, θα δείτε πως είναι πάρα πολύ δύσκολο να χρησιμοποιήσουμε τα κονδύλια, γιατί δεν έχουμε πρόσβαση σε αυτά γιατί χρειάζονται εγγυητές, χρειάζονται εγγυητικές επιστολές, χρειάζεται η κεντρική μας τράπεζα να κάνει τη συζήτηση για το πόσο ε, υπάρχει τρόπος να αναλαμβάνεται ο κίνδυνος αυτός ή να επιδοτείται μέσω κάποιου άλλου χρηματοδοτικού εργαλείου. Τέτοιου είδους συζητήσεις πρέπει να γίνονται όταν λέμε πως χρειαζόμαστε διαφορετικά είδη αναπτυξιακής βοήθειας μέσω εργαλείων που θα μας βοηθήσουν να οικοδομήσουμε το δικό μας δυναμικό με ρεαλιστικό τρόπο. Και τέλος, με πάρα πολλές προσδοκίες αναμένουμε τη συζήτηση για το μελλοντικό πλαίσιο. Γιατί κοιτάξαμε το παρελθόν, το κάναμε σε πολλά ε, βήματα και εσείς και εμείς και είπαμε για να αποτιμήσουμε το πόσο ε, μας ευνόησε το παρελθόν, ποιο ήταν το κόστος που πρέπει να εργαστούμε πιο σκληρά, αλλά για να καταλαβαίνουμε τα θεσμικά πλαίσια όλων, γιατί μιλάει έκθεση και για τη γεωγραφική πραγματικότητα. Εντάξει, μπορούμε αυτό να το δούμε σε φαντασιακό επίπεδο, αλλά θα πρέπει να φτάσουμε και στο σημείο όπου θα συζητάμε ακριβώς τι εννοείται εσείς όταν λέτε γεωγραφικές ιδιομορφίες για το θεσμικό πλαίσιο, το οποίο θα περιγράψει το μέλλον της σχέσης μας. Μια σχέση που επαναλαμβάνω ε, αν υπομονούμε να εγκαθιδρύσουμε. Και σας ευχαριστώ που μου δώσατε το, την ευκαιρία να ε, πάρω το λόγο και να σας μιλήσω. Τα θέματα για τα εργαλεία και τα μέσα είναι μια συνεχιζόμενη συζήτηση στα πλαίσια της αναπτυξιακής βοήθειας που θα γίνει. Επειδή έχουμε καθυστερήσει θα δώσω και σε εσά γρήγορα το λόγο. Είναι η κυρία Χάουτολα. Θα ήθελα να σχολιάσω τα όσα είπε η πρέσβης. Ναι. Κάποιες από τις χώρες της Καρεκόμ, πολλές φορές λόγω τροπικών καταιγίδων για παράδειγμα, α, χάνουν το ΑΕΠ μια χρονιάς ολόκληρης, μέσα σε μια νύχτα. Άρα λοιπόν το θέμα αυτό θα πρέπει να το εξετάσουμε. Ο κύριος Ντούνς. Είπατε πως έχετε καθυστερήσει, οπότε θα προσπαθήσω να είμαι πολύ σύντομος δεν ξέρω πόσο χρόνο έχω στη διάθεσή μου. Καταρχήν να σας ευχαριστήσω και για τα σχόλια και για τις ερωτήσεις που αποδεικνύουν το εξή στα μάτια μου. Πως αυτή τη στιγμή γίνεται ένας λογικός διάλογος που δεν ήταν πάντα ε, ο κανόνας όταν ξεκίνησε ε, ε, όλη αυτή η ιστορία. Γιατί πολλές φορές ε, είχαμε έναν ε, συναισθηματικό, συγκινησιακά φορτισμένο διάλογο για το κατά πόσο χρειάζεται η Συμφωνία Κοτονού κτλ. Χαίρομαι λοιπόν που λόγω των συζητήσεων που έχουμε ήδη κάνει τελικά έχουμε περάσει σε μια συζήτηση που βασίζεται σε επιχειρήματα. Από τις παρεμβάσεις σας καταλαβαίνω πως Πολλές φορές τα επιχειρήματα μας είναι αμυντικά, δηλαδή να μην κάψουμε και τα χλωρά μαζί με τα ξερά. Να δούμε πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα ισχυρά σημεία της συμφωνίας και να τη βελτιώσουμε. Και αυτό ήταν και ο στόχος μας. Και γι' αυτό κάναμε την αξιολόγηση για να δούμε ποιες είναι ε, οι αδυναμίες μας και ποια είναι τα δυνατά μας σημεία. Όχι για να αποδείξουμε ότι δεν λειτουργεί, αλλά για να εντοπίσουμε το πού θα πρέπει να εστιάσουμε τις προσπάθειές μας για να τα πάμε καλύτερα. Το ισχυρότερο συμπέρασμα είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν γίνεται πλήρης χρήση των δυνατοτήτων που προσφέρει αυτή η συμφωνία. Και νομίζω ότι αυτό συμπίπτει σε μεγάλο βαθμό με την προσέγγιση που ακολουθεί ο κύριος Νόιζερ στη δική του γνωμοδότηση. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Θα ήταν πραγματικά πολύ καλύτερο και για εμάς η αξιολόγηση αυτή να έχει γίνει πριν από ένα χρόνο. Ξέρετε όμως κι εσείς πως η προηγούμενη επιτροπή δεν ήταν πολύ δραστήρια στο φάκελο αυτό και χρειάστηκε να γίνουν πάρα πολλές προσπάθειες με πολύ ε, σφιχτές προθεσμίες. Αυτή τη στιγμή προετοιμάζουμε την μετά το κοτονού ε, περίοδο μαζί με την Ευρωπαϊκή Συνένεση, το Consensus, οπότε οι προθεσμίες είναι εξαιρετικά περίπλοκες. Νομίζω όμως πως θα τα καταφέρουμε για κάποια από τα σχόλια α, της συναδέλφου σας για τους τρεις πυλώνες που αποτελούν αυτή τη στιγμή τη βάση της τρέχουσας συμφωνίας, μάλλον θα εγκαταλειφθούν στο μέλλον. Γιατί σε τρεις πυλώνες έχουμε βασίσει κάτι το οποίο ουσιαστικά αποτελεί μια συνεχιζόμενη διαδικασία και που δεν μπορεί κανείς να περιχαρακώσει ή να απομονώσει μια πολιτική ε, για παράδειγμα την εξάλληψη της φτώχειας, εδώ δεν έχει γίνει πλήρης χρήση του δυναμικού ε, που προσφέρεται και εδώ χρειάζεται περισσότερη πρόοδος και για τις τρεις αυτές ε, διαστάσεις. Διαφοροποίηση της οικονομίας. Είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα των όσων σας λέω και όντως έχω αναφερθεί στην αύξηση των εξαγωγών των χωρών και προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και σε ένα μεγαλύτερο μερίδιο των εξαγωγών τους ε, προς τις χώρες μας. Αν όμως αντιστρέψουμε την εικόνα θα δείτε πως όντως είμαστε ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος των χωρών ΑΚΕ και είμαστε ο μεγαλύτερος επενδυτής στις χώρες ΑΚΕ. Και εκεί όμως πρέπει να βελτιωθούμε. Και γι' αυτό προσπαθούμε να βασιστούμε στην ε, συμφωνία ε, οικονομικής εταιρικής σχέσης για να βελτιωθεί το επιχειρηματικό περιβάλλον, το επενδυτικό περιβάλλον και να καταφέρουμε μέσω αυτού να κάνουμε πιο ελκυστικές τις χώρες ΑΚΕ έτσι ώστε να προσελκύουν και εσωτερικές εγχώριες επενδύσεις αλλά και αλλοδαπές επενδύσεις. Και αυτό αποτελεί ένα εκ των ονουκάνευ για τη θεματολογία του Ευρωπαϊκού Κονσένσους και για την κινητοποίηση που πρέπει να γίνει και του εγχώριου ε, εισοδήματος με μεγαλύτερες επενδύσεις από τον εγχώριο ιδιωτικό κλάδο. Μιλήσατε για το γεγονός πως ατενίζουμε υπερβολικά το παρελθόν, το γεγονός πως δεν ε, εξετάζουμε αρκετά το μέλλον. Εμείς το ονομάζουμε επιπτωσιολογική μελέτη όταν γίνεται και έχουμε σχεδόν κλείσει αυτή τη στιγμή. Ε, εξετάζουμε και κάποια ακόμα θέματα κανονιστικά και νομοθετικά. Όμως μόλις είναι έτοιμη αυτή η έκθεση ε, ως έγγραφο εργασίας που θα εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, θα είναι έτοιμο και θα εκδοθεί και θα παρουσιαστεί παράλληλα με την ανακοίνωση του Νοεμβρίου. Και βέβαια θα έχει περισσότερες λεπτομέρειες από την αξιολόγηση όπου θα εξετάσουμε διάφορα σενάρια και εναλλακτικέ λύσεις, θα τα αποτιμήσουμε και μετά θα τα τεκμηριώσουμε έτσι ώστε να έχουμε την τελική ε, επιλογή του προτιμούμενου, ε, της προτιμούμενης εναλλακτικής λύσης που θα πρέπει βέβαια να αποφασίσει ε, το, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Νοέμβριο. Δεν θα είναι ένα νομικό έγγραφο ακόμα με διαπραγματευτική εντολή, Είπαμε πως θα προτιμήσουμε να ξεκινήσουμε με μια ανακοίνωση που είναι πολιτικό έγγραφο που θα περιγράφει όμως την προτιμούμενη επιλογή έτσι ώστε να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε τον πολιτικό διάλογο μαζί σας με τα κράτη-μέλη, με τις χώρες ΑΚΕ και να προετοιμάσουμε καλύτερα το έδαφος για μια πρόταση για διαπραγματευτική εντολή την οποία θα καταθέσουμε ελπίζω μετά το καλοκαίρι του 2017. Τώρα για το τι θα κάνει το Συλλογικό Όργανο των Επιτρόπων, αυτό είναι δικό του θέμα. Δουλεύουμε την ανακοίνωση, θα πρέπει να την τελειώσουμε, να περάσει από τη διοργανική διαβούλευση και βεβαίως την επόμενη εβδομάδα ίσως πρέπει να ρωτήσετε τον Επίτροπο Μίμητσα τι προτιμά. Εγώ ως, ε, αξιωματούχος δεν μπορώ να εκφραστώ αυτή τη στιγμή. Νομίζω όμως πως ξέρετε ε, προς τα που κλείνουμε. Η επιπτωσιολογική μελέτη, θα σχολιάσω το είπε ο κύριος Γκέρεντς, όντως η αξιολόγηση έχει δημοσιευθεί, η επιπτωσιολογική μελέτη και αυτή θα δημοσιοποιηθεί και αναγνωρίζω απολύτως πως θα πρέπει να είναι ε, δημόσιο αυτό το έγγραφο γιατί θα ξεκινήσει μια συζήτηση ε, πάνω σε μια πιο αντικειμενική και πιο σταθερή βάση, κάτι το οποίο δεν συνέβαινε πάντα στο παρελθόν, το είπατε κι εσείς, γιατί είχαμε αποκλίνουσες ερμηνείες κτλ. Οπότε ελπίζω πως το έγγραφο αυτό θα προσφέρει κάτι προς αυτή την κατεύθυνση. Επίσης, συμφωνώ με την ανάλυση που κάνατε για τα ισχυρά σημεία και τα σημεία τα οποία χρήζουν βελτίωσης, όπως επίσης συμφωνώ μαζί σας ε, στην ανάλυση που κάνατε για τα πλεονεκτήματα. Θέλω μόνο να προσθέσω κάτι θα ήθελα να δείτε ολόκληρη την ταινία και όχι μόνο κάποια στιγμιότυπα. Γιατί όταν βλέπουμε μεμονωμένες εικόνες δεν μπορούμε να δούμε το σύνολο. Αν δούμε ολόκληρη την ταινία, όλο το έργο, καταλαβαίνουμε ποια είναι η αρχή και ποιο είναι το τέλος. Από πού ξεκινάμε και πού θέλουμε να φτάσουμε έτσι ώστε να γνωρίζουμε τι μας επέτρεψε να πετύχουμε η Συμφωνία του Κοτονού μαζί με τους εταίρους μας τώρα. Για τη συνεργασία και για τα όσα διακυβεύονται ε, για το συνολικό θεματολόγιο και την παγκόσμια ατζέντα ε, με τον κύριο Γκόμε, που είναι ο συνάδελφο για τι χώρε ΑΚΕ καταλαβαίνω πω υπάρχει ένα εκνευρισμό. παρόλο το δυναμικό, παρόλο το ότι πολύ συχνά όλε οι χώρε, οι 78 των ΑΚΕ έχουν την ίδια άποψη και συμμερίζονται μαζί μα, όταν προσπαθούμε να συνάψουμε μια συμμαχία και να λειτουργήσει όταν ψηφίζουμε σε μια μεγάλη συνδιάσκεψη παγκόσμια δεν είμαστε πάντα πετυχημένοι. Έχουμε παρόλα αυτά ένα καλό παράδειγμα από πέρυσι η COP21 στο Παρίσι, όπου εκεί όντω η συμμαχία λειτουργήσε σωστά και είχαμε και κάποια στιγμή στις διαπραγματεύσεις όπου δείξαμε πως υπάρχει αυτή η πολιτική ε, ηγεσία που δημιουργεί το δυναμικό που χρειάζεται. Για την αξιολόγηση ε, το δείχνει και η επιπτωσιολογική μελέτη. Εδώ ε, έχουμε κάτι που διακυβεύεται, που είναι πώς μπορούμε στο μέλλον να λειτουργήσει αυτή η εταιρική σχέση περισσότερο από ό,τι στο παρελθόν. Και αυτό σχετίζεται και με τους ε, θεσμούς. Εάν καταφέρουμε να εντοπίσουμε τι πράγματι διακυβεύεται και τι, ποιοι είναι οι στόχοι ε, για τους οποίους θα θέλαμε να συνεργαστούμε, ε, σε, για παράδειγμα σε μια τέτοιου είδους παγκόσμια διάσκεψη, τότε θα έχουμε στόχους και όταν έχουμε υπουργικά, κοινά υπουργικά συμβούλια θα μπορούμε να συζητήσουμε τους πραγματικούς στόχους και στις αμυκτές κοινοβουλευτικές συνελεύσεις με θεματολόγιο το οποίο θα είναι ουσιαστικό, σημαντικό γιατί πολλές φορές οι πολιτικοί στόχοι ε, δεν ε, ε, στηρίζονται και από τις χώρες ΑΚΙΑ και από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξίσου. Πρέπει να κάνουμε κάτι παραπάνω στην εταιρική μας σχέση όταν έχουμε θέματα του παγκόσμιου θεματολογίου τα οποία θέλουμε να υπερασπιστούμε. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα από τα πιο σημαντικά σημεία τα, τα οποία θα έπρεπε να μιλήσουμε τώρα για τη δημογραφική πίεση. Είναι ένα θέμα το οποίο αναλύουμε και είναι αρκετά ευαίσθητο σε κάποια σημεία του. Και για να περάσω στο επόμενο σημείο, στα όσα είπε ο κύριος Λίντς για το κατά πόσο νομικά είναι δεσμευτικά τα στοιχεία αυτά. Να πω τα εξή. Είδαμε πως τα όσα είναι νομικά δεσμευτικά στην συνθήκη λειτουργήσαν καλά σε πολλές περιπτώσεις και πως σε άλλες περιπτώσεις δεν επαρκούσαν. Και το καλύτερο παράδειγμα είναι τα ουσιαστικά στοιχεία. Δηλαδή διακυβέρνηση, ανθρώπινα δικαιώματα κτλ. Όπου παρόλο που περιγράφονται σε μια νομικά δεσμευτική συμφωνία, δεν έχουν επαρκέσει για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός. Και γι' αυτό ίσως θα έπρεπε να το έχουμε διατυπώσει κάπως διαφορετικά, δηλαδή να μην λέμε πως... Ε, δεν πετύχαμε ε, τα πάντα στα νομικά δεσμευτικά σημεία, θα έπρεπε να πούμε ότι ίσως δεν επαρκεί ο τρόπος αυτός. Για τα όσα είπε η κυρία Χάουτο, αλλά και για τη διαφάνεια, ε, την ε, κοινωνία των πολιτών, τις γυναίκες, τη λογοδοσία. Συμφωνώ και για τόσο από ο κύριος Γκέρν σε σχέση με το παρελθόν προοδεύσαμε. Αλλά προφανέστατα μια αξιολόγηση και ένα έγγραφο στο μέλλον που θα περιγράφει την κατάσταση και όπου θα λέμε πως χρειάζεται περισσότερη πρόοδο στο μέλλον με ε, πιο στεναρό ρόλο για τα εθνικά κοινοβούλια, για την ε, κοινωνία των πολιτών, για τον ιδιωτικό κλάδο ε, χρειάζεται. Και στη διαβούλευση που έχουμε κάνει δείχνει πως επί χάρτου και στην πραγματικότητα τα πράγματα έχουν προοδεύσει, αλλά υπάρχει σαφέστατα περιθώριο για μεγαλύτερη πρόοδο και σε μια μελλοντική εταιρική σχέση θα πρέπει στα σημεία αυτά να πάμε πιο κάτω στην γνωμοδότηση που θα εγκρίνεται σήμερα το απόγευμα, νομίζω ότι η ορολογία που χρησιμοποιείται και η διατύπωση συμπίπτουν σε πολύ μεγάλο βαθμό με τις δικές μας σκέψεις. Και τα όσα είπε ο κύριος Βέντα και το πώς ε, σχετίζεται με τα SDG, νομίζω πως εδώ έχουμε το πλαίσιο έχουμε τον τρόπο με τον οποίο θα μεταφερθούν αυτά στην αναπτυξιακή βοήθεια μέσω του Ευρωπαϊκού Κονσένσους και έχουμε και τα γεωγραφικά ε, στοιχεία για τις 78 χώρες ΑΚΕ, τα οποία θα ληφθούν υπόψη έτσι όλα αυτά να εφαρμοστούν ε, με το σωστό τρόπο στην μετά εποχή. Κυρία Πρόεδρος, σειράξεις ασφάλεια συμφωνώ απόλυτα. Η συνολική στρατηγική που παρουσιάσαμε καλύπτει τα θέματα αυτά και περάσαμε από τις διακρατικές σειράξεις στις ενδοκρατικές σειράξεις. Έχουμε μια τελείως διαφορετική εικόνα που δεν συμπίπτει με την ε, παλαιότερη ανάλυση που κάναμε. Έχει εντάξει μια νέα διάσταση. Έχουμε τη ριζοσπαστικοποίηση και βλέπουμε την Ιγυρία, την Πόκο Χαράμ, τη Σομαλία, την Αλσαμπάπ και πολύ καλά τέτοια παραδείγματα. Άρα λοιπόν αυτό το νέο μοντέλο σειράξεων έχει ήδη ενταχθεί στο μοντέλο σκέψης και θα αποτελέσει κομμάτι αναπόσπαστο οποιασδήποτε συζήτηση για τη μετά του Κοτονού συμφωνία. Για την ευελιξία της ε, χρηματοδότησης συμφωνώ μαζί σας. Και για μας πολλές φορές είναι πολύ δύσκολο το γεγονός ότι έχουν κλειδωθεί σε πολυετή προγράμματα τα κονδύλια και δεν είναι εύκολο πάντα να είναι πιο ευέλικτη η χρηματοδότηση. Η αξιολόγηση αποδεικνύει πως όμως αυτή η μακροπρόθεσμη σταθερότητα και στόχευση προσφέρει και πλέον εκτήματα. Γιατί δηλαδή παραμένουμε ε, στη σωστή πορεία και αποφεύγουμε από χρόνο σε χρόνο να ε, παραπέουν κονδύλια προς τη μία ή προς την άλλη κατεύθυνση αναλόγως και με την τραγωδία που είναι στην επικαιρότητα. Τώρα, αν δεν κανείς τώρα την, το προσφυγικό, ναι, είναι ένα νέο πολιτικό θέμα στην κορυφή του θεματολογίου και προσπαθούμε να δούμε πόσο μέσω αντιξιακής βοήθειας μπορούμε να προσφέρουμε. Αυτό δεν έρχεται απαραίτητα σε σύγκρουση με τα κονδύλια τα οποία έχουν ήδη προγραμματιστεί, γιατί αυτό που κάναμε τελικά με το θέμα της φτώχειας και με το θεματολόγιο ε, για τις αλλαγές που θέλαμε να εισάγουμε, ε, νομίζω ότι ανταποκρίνεται στα όσα θα έπρεπε να κάνουμε για να εξαλειφθούν οι ρίζες ε, του κακού. Άρα λοιπόν δεν χρειάζεται μία, α, έναν απόλυτο επαναπρογραμματισμό, αλλά στα πλαίσια της αναθεώρησης που θα γίνει θα κάνουμε κάποιες προσαρμογές. Όμως χρειαζόμαστε περισσότερη ευελιξία για να καταλήξουμε σε ένα σύστημα το οποίο θα συμφωνήσουμε όλοι και που θα αποτελεί ένα από τα πλέγματα των θεμάτων που αντιμετωπίζουμε ε, για τη μετά το Κοτονού Συμφωνία. Την ερώτηση του κυρίου Πρέντα, βεβαίως, για τους συνολικούς στόχους ανάπτυξης, βεβαίως, οπωσδήποτε, θα λάβουμε υπόψη την ε, κατάληξη της Ευρωπαϊκής Συνενετικής ε, Στάσης για τους βιώσιμους αναπτυξιακούς στόχους SDG και βεβαίως ε, και αν κάνουμε μια αποτίμηση του τι κάνουμε είμαστε στην πρωτοπορία αλλά φυσικά μπορούμε να κάνουμε περισσότερο και όπου μπορούμε θα το κάνουμε. Νομίζω ότι ε, για τον περιορισμένο χρόνο που είχα προσπάθησα να τα αντιμετωπίσω όλα. Πρόεδρος, ευχαριστώ για την ε, πολύ αναλυτική αντιμετώπιση σας, για το ότι απαντήσατε σε όλες τις ερωτήσεις. Βοηθάει τη συζήτησή μας, όχι μόνο για την κατάσταση του μετά την Συμφωνία Κοτονού, αλλά και το πώς θα διαμορφώσουμε συνένεση και για το επόμενο θέμα που είναι η αποτελεσματικότητα της ε, αναπτυξιακής βοήθησης. Ευχαριστούμε τον κύριο Ντούνς που ήρθε και ήταν πάντα ιδιαίτερα επικοδομητικός. Όπως πάντα η Επιτροπή Ευχαριστώ. Ωραία, θα ψηφίσουμε σήμερα το απόγευμα την έκθεση του κυρίου Νόιζα. Λοιπόν, άρα πολύ εύκολα περνάμε στο επόμενο θέμα, αύξηση της ε, αποτελεσματικότητα, της αναπτυξιακή βοήθειας. Παρακαλώ όσοι φεύγουν να μην θορυβούν. Είναι λοιπόν το 5, αύξηση της αποτελεσματικότητα τη αναπτυξιακή συνεργασία θα προετοιμάσουμε μια έκθεση πρωτοβουλία για το θέμα αυτό. Ο εισηγητής θα είναι ο κ. Πρέντα, που είναι ο μόνιμος εισηγητής μας για τα θέματα αυτά. Υπάρχει μια πολύ σημαντική συνδιάσκεψη στο Ναϊρόμπι αργότερα φέτος, 28 Νοεμβρίου με 1 Δεκεμβρίου. Στη διάσκεψη αυτή θα συνεχίσουμε την εργασία προηγούμενων προσπαθειών. Να σας δώσω ένα πλαίσιο για να σας βοηθήσω να καταλάβετε γιατί συζητάμε το θέμα αυτό της αποτελεσματικότητας της αναπτυξιακής βοήθειας. Το 2005 η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι κυβερνήσεις ενέκριναν την δήλωση των Παρισίων για την αποτελεσματικότητα της βοήθειας που τόνισε ότι υπάρχουν πέντε θέματα, η αποδοχή από τη χώρα, η ε, εναρμόνιση με την ε, κατάσταση της χώρας και η ε, κοινή λογοδοσία. Αυτά έγιναν το 2005-2008 στην Ακρά, ξανασυναντήθηκαν οι κυβερνήσεις και συμφώνησαν ότι τα θέματα των Παρισίων ήταν σωστά, αλλά έπρεπε να γίνουν περισσότερα για να είναι αποδεκτά τα προγράμματα αυτά από τις χώρες, ε, να συμμετέχουν περισσότεροι στην ψυχική συνεργασία, δηλαδή η ΜΚΟ και τα κοινοβούλια, να είναι μετρήσιμα τα αποτελέσματα και να βελτιώσουμε τη δυνατότητα των χωρών να ε, διαχειριστούν την ανάπτυξή τους. Και πρόσφατα, πριν από πέντε χρόνια, στο Μπουσάν υπήρξε ένα φόρουμ υψηλού επίπεδου το Δεκέμβριο του 2011 με αποτέλεσμα τη δημιουργία της ε, παγκόσμιας εταιρικής σχέσης για την ανάπτυξη της συνεργασίας, να περάσουμε από την έμφαση στην αποτελεσματικότητα της βοήθειας στο ευρύτερο θέμα της αποτελεσματικής ανάπτυξης. Ο κύριος Πρέντα νομίζω ήταν ο εισηγητής μας τότε το 2011 για το θέμα αυτό. Τώρα λοιπόν Προετοιμάζουμε την επόμενη σημαντική διεθνή συνδιάσκεψη. Έχουμε δύο προσκεκλημένου ομιλητέ, Η πρώτη είναι Ναντίν Κεμπόσο, που είναι ε, στο τμήμα τη ε, Παγκόσμια Ανάπτυξη συνεργασία του ΟΟΣΑ και από ό,τι κατάλαβα εκπονεί ο ΟΣΑ μια έκθεση για την περισσότερη αποτελεσματικότητα της αναπτυξιακής συνεργασίας. Είστε λοιπόν βασικό ομιλητής ε. και επίσης είναι εδώ και η Σουζάννα Σκλατκόβα από το Concord που προσπαθεί να αυξήσει την ε, ε, αποτελεσματικότητα της βοήθειας. Και έχουμε και ε, συναδέλφους από την Γενική Διεύθυνση Ντεύκο που θα μιλήσουν αργότερα. Αλλά δεν ξέρω εάν πριν τους ομιλητές θέλει να πει τίποτα ο κύριος Πρέντα. Όχι, θα μιλήσει μετά. Ωραία, να ακούσουμε πρώτα τους προσκεκλημένους μας. Όπως σας είπα, εκπονούμε μια έκθεση πρωτοβουλίας για το θέμα αυτό που ε, θα μας απασχολήσει πριν από την διάσκεψη στο Ναϊρόμπι είναι σημαντικό για τη διαμόρφωση της νέας συνένεσης για την μετακοτονού κατάσταση και την εφαρμογή των STG, των βιώσιμων αναπτυξιακών στόχων. Παρακαλώ, έχετε το λόγο, κυρία Γκμπόσα. Βεβαίω, είμαι από τον ΟΣΑ, λέει κυρία Γκμπόσα, και όπω γνωρίζετε, ο ΟΣΑ μαζί με το UNDP είναι οργανισμός που προσπαθεί να προωθήσει τα θέματα της αποτελεσματικής αναπτυξιακή συνεργασίας. Ξέρετε τι σημαντικές εξελίξεις έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια γι' αυτό, αλλά να υπενθυμίσω μερικά θέματα που έχουν να κάνουν ειδικά με την αναπτυξιακή συνεργασία, η οποία έχει αλλάξει ριζικά, όπως ξέρετε, τις τελευταίες δεκαετίες. Η σημασία της βοήθειας έχει μειωθεί, δηλαδή το ύψος ε, σε σχέση με ιδιωτικούς πόρους και εγχώρους πόρους, αλλά συμμετέχουμε στη διαχείρισή της. Όσο ΩΣΑ και το 2015 συνεχίζουμε να διαπιστώνουμε ότι η αναπτυξική βοήθεια είναι ο σημαντικότερος εξωτερικός πόρος για την ανάπτυξη. Κάτι άλλο σημαντικό είναι ότι οι πηγές της αναπτυξιακής ε, επιδότησης έχει αυξηθεί ο ρόλος ε, των φιλανθρωπικών πόρων, ε, ιδιωτικοί πόροι και μη καπαόμικρον συμμετέχουν και αυτοί στη χρηματοδότηση. Αυτές οι εξελίξεις κατέληξαν στην διακήρυξη του Μπουζάν και για να καταλαβαίνουμε τι λέμε, η διακήρυξη αυτή υπεγράφει το 2011 με στόχο να συμμετέχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι, όχι μόνο οι κυβερνήσεις όπως το Παρίσι, αλλά να συμμετέχουν και όλοι οι άλλοι εμπλεκόμενοι, ιδιωτικό τομέα, η κοινωνία των πολιτών, οι φιλανθρωπικοί φορείς και άλλοι ε, χρηματοδότες, ούτως ώστε να συνεργάζονται όλοι με βάση τα πλεονεκτήματα του καθενός. Για παράδειγμα, το πλεονόκτημα, τα πλεονεκτήματα των ιδιωτικών φορέων ε, δεν είναι τα ίδια με τα πλεονεκτήματα των κυβερνήσεων ή φορέων της κοινωνίας των πολιτών. Η διακήρυξη του Μπουζάν οδήγησε στη συμφωνία ή τις αρχές του Μπουζάν, που είναι εξέλιξη της ε, δήλωσης των Παρισίων, και βασίζεται σε πέντε αρχές. Πρώτα απ' όλα αποδοχή, συντονισμός με τις προτεραιότητες της χώρας, εστίαση στα αποτελέσματα, δέσμευση για διαφάνεια και λογοδοσία για τους πόρους για την ανάπτυξη και ένα νέο στοιχείο η δήλωση για να υπάρξουν εταιρικέ σχέσεις ε, με συμμετοχή ευρύτερη για να υπάρξει και καλύτερο αποτέλεσμα. Ένα άλλο σημαντικό αποτέλεσμα από τη συνάντηση του Μπουζάν είναι η δημιουργία της παγκόσμιας εταιρικής σχέσης για αποτελεσματική αναπτυξιακή συνεργασία. Και τι είναι αυτό, ρωτάνε πολλοί, είναι ένα σώμα που έχει στόχο να επιτηρεί την αποτελεσματικότητα της αναπτυξιακής συνεργασίας, όπου συμμετέχουν σε τακτικές συναντήσεις εκπρόσωποι της αναπτυξιακής κοινότητας για να δούμε πώς θα πάμε, πού έχει υπάρξει πρόοδος, που υπάρχουν προκλήσεις, τι περισσότερο μπορούμε να κάνουμε για να έχουμε καλύτερο αποτέλεσμα. Για να το κάνει αυτό, αυτή η παγκόσμια εταιρική σχέση έχει δημιουργήσει ένα πλαίσιο επιτήρησης με βάση 10 δείκτες για να δούμε πώς θα πάνε όσοι συμμετέχουν στην παροχή και διαχείριση αναπτυξιακής βοήθειας. Πώς θα πάει ο προπολογισμό βασίζονται στις δυνατότητε της χώρας, βασίζονται στους στόχους της χώρας, αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί αυτό το πλαίσιο επιτήρησης μας παρέχει στοιχεία και αριθμούς και δεδομένα που παρουσιάζονται στην αναπτυξιακή κοινότητα τακτικά για να δούμε πώς θα πάμε, αλλά και για να προωθήσουμε αυτό που αποκαλούμε αμοιβαία λογοδοσία. Είναι διάλογος μεταξύ αναπτυσσόμενων και αναπτυγμένων χωρών, όλων των εμπλεκόμενων φορέων, για να δούμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την προσπάθειά μας, που επιτυγχάνουμε τους στόχους μας και που όχι. Στα πλαίσια της, ε, του θεματολογίου 2020 έχει τεθεί το ερώτημα αυτές οι αρχές εξακολουθούν, είναι σημαντικές. Είπατε ότι θα γίνει στο Αερόβι μια συζήτηση υψηλού επίπεδου τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο, όπου θα συναντηθούν οι εμπλεκόμενοι φορείς για να δούνε πόσο αποτελεσματική είναι η συνεργασία τους για την ανάπτυξη. Άρα το ερώτημα είναι θα κάνουμε άλλη μια μεγάλη συνάντηση χωρίς πολύ αποτέλεσμα ή αν θα είναι σημαντική θα έχει αποτελέσματα. Και θα σας εξηγήσουμε γιατί θεωρούμε ότι έχουμε κρίσιμα θέματα ενώπιόν μας. Γιατί λοιπόν αυτή η συνάντηση στο Ναϊρόμπι είναι σημαντική για όλους τους εμπλεκόμενους και πρέπει να παρευρεθούν όλοι. Πρώτον, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΣΑ έκανε μια παρομοίωση. Όλοι μιλάμε για την πλοήγηση με δορυφόρους, GPS. Ε, θα παρομοίαζα την προσπάθειά μας με το GPS της αναπτυξιακής συνεργασίας. Σου λέει πού να πας και πώς να φτάσεις. Είναι σημαντικό να έχεις στόχους. Γιατί καθορίζοντας στόχους, πιέζουμε τις κυβερνήσεις, τους εμπλεκόμενους, να επιδείξουν ότι επινηχάνουν πρόοδο. Γιατί μπορούν οι εκλογείς τους, οι συνεργάτες τους, οι εταίροι τους να δουν σε τι βαθμό έχουν επιτύχει τους στόχους τους. Έτσι ε, δημιουργούμε και το πλαίσιο για τη λογοδοσία. Οι αναπτυσσόμενες και οι ανεπτυγμένες χώρες πρέπει να λογοδοτήσουν με βάση αυτές τις αρχές αυτό το πλαίσιο. Και η συνάντηση θα είναι μια δυνατότητα να κάνουμε διάλογο υψηλού επίπεδου, να δούμε πού πρέπει να κάνουμε περισσότερα, πού πρέπει να τα πάμε καλύτερα. Και αυτό συνήθως οδηγεί στην ανάληψη δεσμεύσεων. Και ξέρουμε ότι τα SDG και τα NDG ήταν δεσμεύσεις που αφορούσαν την αναπτυξιακή συνεργασία. Στον Αερόμπι αυτές οι δεσμεύσεις, ούτω ώστε να γίνει πιο αποτελεσματική η συνεργασία και να επιτευχθούν οι στόχοι SDG, εκεί θα συζητηθεί αυτή η προσπάθεια. Είναι σημαντικό να συζητηθούν οι στόχοι αυτοί, γιατί η εφαρμογή τους είναι ουσιώδης και μπορεί να γίνει μόνο μέσω συνεργασίας. Γι' αυτό πρέπει και εσείς να πάτε στον Αερόμπι. Μία άλλη ερώτηση που μου ζητήθηκε να ε, σας αναφέρω είναι πόσο επιτυγχάνουμε τους στόχους. Πόση πρόοδο επιτυγχάνουμε. Αυτό το παγκόσμιο πλαίσιο εταιρικής σχέσης συζητάει κάθε δύο χρόνια πώς θα πάει η αναπτυξιακή συνεργασία και πιστεύω ότι έχει υπάρξει πραγματική αύξηση της αποτελεσματικότητας. Οι συναντήσεις επιτήρησης δείχνουν ότι υπάρχει διαρθρωτική αλλαγή στη συμπεριφορά των εμπλεκομένων. Πρώτα απ' όλα υπάρχει ένα πλαίσιο αποτελεσμάτων με το οποίο μπορούν να μετρήσουν όλοι οι εμπλεκόμενοι. Και επίσης έχουν προσαρμόσει τη δράση τους στην ε, πολιτική και στους στόχους και τις μεθόδους της χώρας. Και έτσι, οπωσδήποτε, έχουμε ένα μέτρο αποτελεσματικότητας. Γιατί η διαφάνεια τώρα και την προβλεψιμότητα της χρηματοδότησης ανάπτυξης. ή γύρια αυτή επέδειξαν επέδειξαν ότι πάνω από 80% της βοήθειας τώρα βασίζεται σε αυτήν την προβλεψιμότητα δίδεται για συγκεκριμένους στόχους που πρέπει να επιτευχθούν κάθε οικονομικό έτος. Βεβαίως, όλοι δεν έχουν ακόμη κάθε πληροφόρηση και ιδίως οι χώρες, αλλά έχει υπάρξει πρόοδος. Όπως σας είπα, το 80% δεν συνδέεται με όρους, για παράδειγμα, όσον αφορά τους προμηθευτές και όλοι οι εμπλεκόμενοι συμμετέχουν στην ε, προσπάθεια να υπάρξει και να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον που να βοηθάει τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών και του ιδιωτικού τομέα. Έτσι λοιπόν το θεματολόγιο και οι στόχοι αποτελεσματικότητας είναι ποιοτικό άλμα για να πιέσουν και τις αναπτυγμένες και τις αναπτυσσόμενες χώρες να επιτύχουν τους κοινού τους στόχους. Προφανές φαίνεται να είναι αποδεκτή η στόχη από τη χώρα που λαμβάνει τη βοήθεια, αλλά δεν είναι πάντα προφανής η επίτευξη αυτού του στόχου. Παρ' αυτά έχει υπάρξει πρόοδος. Αυτό σημαίνει ότι το θεματολόγιο το 2030 δεν θα, υπάρξει, δεν θα δημιουργήσει προβλήματα για την υιοθέτησή του στον αερόμπι. Μπορείτε να φανταστείτε ότι το θεματολόγιο του 2020 ε, είναι ένα θεματολόγιο που προσπαθεί να αλλάξει την κατάσταση, άρα θα έχει επιπτώσεις. Ποιες θα είναι. Πρώτα απ' όλα, οι δεσμεύσει που ήδη ανέφερα. Η επίτευξη αυτών των δεσμεύσεων τα αποτελέσματα του 2016 ακόμη τα μελετάει ο ΩΣΑ και θα σας τα πούμε στον αερόμπι αλλά μπορώ ήδη να σας πω ότι σε γενικές γραμμές θα πάμε καλά. Νομίζω ότι θα φτάσουμε σε αποδεκτό επίπεδο σε σχέση με το στόχο που είχαμε προκαθορίσει. Αλλά έχει υπάρξει κάποια στασιμότητα. Για τους περισσότερους ε, στόχους έχουμε επιτύχει ποσοστά 75-80% αλλά τα τελευταία χρόνια δεν έχει υπάρξει επαρκής πρόοδος. Πρέπει να δούμε λοιπόν αν υπάρχουν κάποιοι, κάποιοι δομικοί, διαθροτικοί φραγμοί, γιατί υπάρχουν. Πρέπει λοιπόν να γίνει κάτι για αυτούς. Και αυτό ορισμένοι εμπλεκόμενοι το αποκαλούν ε, στόχοι ανεκπλήρωτοι ακόμη. Πρέπει να καταλάβουμε ότι έχουμε φτάσει σε ένα κάποιο επίπεδο, τώρα πρέπει να ανέβουμε στο επόμενο επίπεδο. Πρέπει λοιπόν να αυξήσουμε και την επίπτωση της αναπτυξιακής συνεργασίας. Και πρέπει λοιπόν στον Αερόμπι να συζητήσουμε πώς θα το κάνουμε. Δεύτερη πρόκληση για τον Αερόμπι. Όσο εξετάζουμε αυτή την αρχή, καταλαβαίνουμε ότι κυρίως αφορούν τους δημόσιους φορείς που ασχολούνται με την αναπτυξιακή βοήθεια. Είναι δύσκολο να επιβάλλουμε σε ιδιωτικού φορείς τέτοιους στόχους. Αλλά στο Μπουζάν δηλώσαμε ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι πρέπει να ασχοληθούν με βάση το συγκριτικό πλεονέκτημα του καθενός. Άρα ένα σημαντικό θέμα είναι πώς μπορούμε να έχουμε την πλήρη δέσμευση και του ιδιωτικού τομέα. Ξέρουμε ότι η χρηματοδότηση SDG δεν θα επιτευχθεί εάν δεν υπάρξει και ιδιωτική χρηματοδότηση. Αυτό είναι το βασικό μας καθήκον για την επόμενη περίοδο. Και έχουμε μελέτες που δείχνουν ότι η δέσμευση των ε, ιδιωτικών φορέων για τους στόχους SDG είναι ακόμη περιορισμένη. Πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να υπάρξει περισσότερη ιδιωτική χρηματοδότηση. Έχουμε πολλά επιτυχημένα παραδείγματα πώς μπορούμε να βοηθήσουμε, για παράδειγμα, μειώνοντας ε, τους κινδύνους για τον ιδιωτικό τομέα ε, σε τομείς που δεν είναι ε, εύκολα επικερδής ή μέσω εταιρικών σχέσεων μεταξύ δημοσίων και ιδιωτικών φορέων. Πώς μπορούν λοιπόν οι δυνατότητές μας να αυξήσουν τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα γιατί όπως καταλαβαίνετε, όπως ήδη σας είπα, οι ιδιωτικοί φορείς δεν είναι οι πιο προσαρμοσμένοι για ορισμένους από τους στόχους μας. Επίσης, θέλουμε να συμβάλλουμε στη διαδικασία παρακολούθησης και συνέχισης από πλευράς του ΟΗΕ που μετράει πώς θα πάνε όλοι οι εμπλεκόμενοι. Θέλουμε οπωσδήποτε να έχουμε αρκετά στοιχεία που να είναι στη διάθεση της διεθνούς κοινότητας για να μπορούμε να μετρήσουμε την ε, αποτελεσματικότητα της βοήθειας, πώς μπορούμε να ε, ε, αντλήσουμε περισσότερους πόρους από την κοινωνία των πολιτών και τον ιδιωτικό τομέα. Στον αερόμπι λοιπόν θα εξεταστούν αναλυτικά τα θέματα αυτά με συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων για να δούμε πώς θα πάμε, πού πρέπει να γίνουν σοβαρές αλλαγές και ελπίζω να υπάρξει συμμετοχή υψηλωτά του επίπεδου από τις κυβερνήσεις, τον ιδιωτικό τομέα και να οδηγήσει σε νέες δεσμεύσεις για να εργαστούμε στους τομείς που προανέφερα, ούτω ώστε βασικά να προσαρμοστεί η συνεργασία στο επίπεδο των θεμάτων που αντιμετωπίζουμε. Σας ευχαριστώ, λέει η κυρία Μακάβαν, που συνδέσατε το θέμα αυτό με τα ευρύτερα θέματα. Είναι πολύ σημαντικό για να καταλάβουμε πώς συνδυάζονται όλες αυτές οι διεθνείς συνδιασκέψεις. Και τώρα η Σουζάννα Σλακόβα από τον οργάνωση Κόγκορτ. Πείτε μας ε, τι κάνει η κοινωνία των πολιτών. Ε, Εμείς ε, είμαστε μια πλατφόρμα η οποία ε, στην οποία συμμετέχουν πολλές μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Δουλεύουμε βέβαια πολύ στενά ε, ε, και από το, την, Παρίσι στην παγκόσμια συνεργασία μέσω της πλατφόρμας που ονομάζεται Συνολική Συνεργασία για την Καλύτερη Αποτελεσματικότητα. Είμαστε δύο χρόνια πριν το Μεξικό και ήρθαμε εδώ έτσι ώστε να σας κάνουμε μία αποτίμηση όσον αφορά την πρώτη μας ε, φάση εργασίας. Ε, θα πρέπει εδώ, θέλω να σας πω τι έγινε ε, στο Μεξικό ή μάλλον τι κάναμε από το Μεξικό. Θα θυμάστε ότι το θέμα της αποτελεσματικότητας ήταν ένα από τα κεντρικά ζητήματα της διάσκεψης για τη χρηματοδότηση αλλά και τη διάσκεψη κορυφής για τους ανεπτυξιακούς στόχους SDGs. Οι βασικές αρχές έχουν έχουν ε, ε, καθοριστεί και ε, βεβαίως έχουν έχουν οριστεί ε, και ο ρόλος των κατευθυντηρίων αρχών των Ηνωμένων Εθνών. Ε, σαν Concord θεωρούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχασε ε, την ευκαιρία να δημιουργήσει κάποιους συνολικούς στόχους για την αναπτυξιακή αποτελεσματικότητα. Είναι γεγονός ότι υπάρχει μια παλαιά εμπειρία, αλλά η διαφάνεια, ο η απόδοση ευθυνών ε, και ε, όλες οι υπόλοιπες αρχές οι οποίες σχετίζονται με τη λογοδοσία ε, πρέπει να είχαν βασιστεί περισσότερο σε αυτές τις οχτώ βασικές τάσεις. Τι ε, εννοούμε με αυτό. Θέλουμε η συνεργασία, η αναπτυξιακή βοήθεια να είναι καλά ε, συντονισμένη και βεβαίω να έχει σχεδιαστεί από τους ίδιους τους πολίτες των αναπτυσσόμενων χωρών. Ε, αυτό αποτελεί σημαντικό διακύβευμα έτσι ώστε για τις νέες, έτσι ώστε το νέο χρηματοδοτικό τοπίο να είναι πιο αποτελεσματικό. Πρόκειται για μια καλή ευκαιρία να μπορέσουμε να χτίσουμε, να οικοδομήσουμε πάνω στις παλαιές ε, συνεργασίες, ε, πάνω σε αυτές τις ατελείς ονομαζόμενες εργασίες ε, του Παρισιού, έτσι ώστε να τις ολοκληρώσουμε και βεβαίως να έχουμε καλύτερη υλοποίηση όλων αυτών των αρχών. δεν υπάρχει άλλος καλύτερος τρόπος επιτήρησης monitoring ε, από την συμμετοχή πολλών ε, εμπλεκομένων. Θα πρέπει να μην ε, λησμονούμε και τον λόγο για τον οποίο έχουν δημιουργηθεί αυτές οι κατευθυντήριες αρχές οι οποίες αναφέρονται και στη Συμφωνία του Μπουζάνα. Δηλαδή κυρίως δημιουργήθηκαν έτσι ώστε να υλοποιηθούν οι πολιτικές διασμεύσεις και και ε, ε, οπωσδήποτε δεν θα πρέπει να ε, αποβούν οι αρχές αυτές σε ζημία των αρχών λογοδοσίας. Έλεγα λοιπόν ότι αυτή είναι μια καλή ευκαιρία έτσι ώστε να επιτύχουμε τους στόχους, αλλά όχι μόνο αυτό. Θα πρέπει να βασίζονται σε σωστή και αντικειμενική και ανάλυση ε, στοιχείων. Ε, οι μεμονωμένες χώρες ε, θα πρέπει να αναλάβουν διορθωτικές δράσεις έτσι ώστε να ξαναμπούν στην σωστή τροχιά. Οι τάσεις της αναπτυξιακής συνοχής είναι σημαντικές, γι' αυτό λοιπόν έχουμε εκδώσει την τελευταία ετήσια έκδοση. Κάνουμε τέτοιες εκδόσεις τα τελευταία 11 χρόνια έτσι ώστε να μπορούμε να παρακολουθήσουμε την τροχιά των θεμάτων αυτών. Θα σας πω και δύο στοιχεία τα οποία θα περιλαμβάνονται και στην ανάλυση ε, αυτού του έτους. Θα αναφερθεί ότι ε, τα περισσότερα, οι περισσότερες χώρες ε, αντιμετωπίζουν ως δεσμευτικές τις συμφωνίες Άκρα και Παρισίων, αλλά δεν υπάρχει ακόμα αρκετός χρόνος έτσι ώστε μέχρι τον Μπουζάν να έχουν προχωρήσει κάποιες καταστάσεις. Εμείς θέλουμε να συμπεριληφθούν οι βασικές αρχές της ανάπτυξης στα αναπτυξιακά προγράμματα, περισσότερο από όσο γίνεται μέχρι τώρα η Γερμανία ε, έχει ε, ε, ένα, συγκεκριμένο τμήμα όσον αφορά την αποτελεσματικότητα της αναπτυξιακής βοήθειας. Η Ρουμανία, η Ιταλία επίσης έχουν εντάξει ένα τέτοιο τμήμα και μια τέτοια αναφορά στον αναπτυξιακό νόμο, αλλά ας πούμε η Ιταλία έχει ένα εθνικό πολυμερές συμβούλιο το οποίο εργάζεται ακριβώς επί θέματος τη συνοχή στρατιωτικής βοήθειας. Ε, το Λουξεμβούργο ε, ε, διαθέτει ένα σχέδιο δράση όσον αφορά την αποτελεσματικότητα, αλλά στην Σλοβακία και την Ισπανία απλώ περιλαμβάνονται κάποιε αρχέ αποτελεσματικότητα στα βασικά του αναπτυξιακά προγράμματα. Το πρόβλημα γενικότερα είναι ότι οι περισσότερε ευρωπαϊκέ χώρε ναι, έχουν προοδεύσει όσον αφορά τις κοινέ στρατηγικές Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, όσον αφορά δηλαδή τις αρχές που είχαν καθοριστεί στο Μεξικό, αλλά δυστυχώς αυτό που βλέπουμε ε, είναι ότι οι 13 ε, χώρες κυρίως της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν δώσει πρωταρχικότερο ρόλο στον ιδιωτικό τομέα εν ώψη και του Ναϊρόμπι και της διάσκεψης αυτής. Να υπενθυμίσω ότι οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών δεν έχουν και τις ίδιες ευκαιρίες σε ολόκληρο τον κόσμο. Ε, γιατί υπάρχουν ανοίγματα παντού ε, προς τον ιδιωτικό ε, τομέα. Ε, φαίνεται πάντως ότι ε, δίνεται περισσότερη σημασία στον ιδιωτικό τομέα παρά στη λογοδοσία και την ε, διαφάνεια. Εμείς θεωρούμε ότι θα πρέπει να υλοποιηθούν ή τα, συμφωνηθέντα σε διεθνές επίπεδο, κυρίως όσον αφορά τις βασικές αρχές. Αυτό που περιμένουμε εμείς και προσδοκούμε σαν Concord από το Ναϊρόμπι είναι το εξής. Μάλλον πριν από τη συνεδρίαση του Ναϊρόμπι ε, ε, θα θέλαμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να ε, έχει μια φιλόδοξη κοινή θέση η οποία θα διασφαλίσει κάποια πρόοδο όσον αφορά την συνολική συνεργασία. Αυτό δεν μπορεί να γίνει όμως εάν δεν υπάρξει και ταυτόχρονα δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα βάσει και της διάσκεψης της άκρα θα πρέπει να ε, ε, ισχυροποιηθούν ε, οι αρχές του, στο Μπουζάν και επίσης θα πρέπει να υπάρξουν και εκθέσεις πρόοδου σε σχέση με τις αρχές του Μπουζάν με τρόπο ώστε να μπορέσουν να υλοποιηθούν σε τακτική βάση οι αρχές του Μπουζάν με τακτική επιτήρηση και έκθεση ανά 24 τουλάχιστον μήνες. Ε, επίσης ε, και τα Ηνωμένα Έθνη, ε, ο τομέας των βασικών κατευθυντηρίων αρχών, θα πρέπει να επιτηρεί την όλη κατάσταση, έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι ότι οι δεσμεύσεις και οι αρχές του Μπουζάν μπορούν και πρέπει να υλοποιηθούν. Να υπενθυμίσω για μία ακόμα φορά ότι ε, το πρόγραμμα ε, επιτήρησης ε, περιλαμβάνει και την κοινωνία των πολιτών, ενισχύει την αμοιβαία λογοδοσία και προωθεί τον διάλογο μεταξύ των αναπτυσσομένων εταίρων. Φρονούμε ότι είναι σημαντικό ε, ε, να ε, υπάρξει συγκεκριμένη αναφορά στα αποτελέσματα του GPDC καθώς επίσης και τις εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την υλοποίηση και προώθηση των αρχών της αποτελεσματικότητας της αναπτυξιακής βοήθειας. Και είμαστε εδώ για να ζητήσουμε από εσά, από τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, να ζητήσουν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να οργανώσει σε ευνοσιακό επίπεδο έναν πολυμερή διάλογο και ανταλλαγή απόψεων πριν, τον, πριν το ε, Ναϊρόμπι. Και επίσης ε, να σας πω ότι στις 26 Οκτωβρίου θα έχουμε και την ε, δημοσιοποίηση της έκθεσής μας ένα μήνα σχεδόν πριν από τον Ναϊρόμπι. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε πρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην οποία θα δώσουμε το λόγο λίγο αργότερα. Θα δώσω τώρα το λόγο πρώτα στον κύριο Πρόεδρε και μετά σε όσους συνάδελφους ζήτησαν το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε πολύ και τις ε, κυρίες ε, για τις ε, παρεμβάσεις που έκαναν. Θα ήθελα να πω, να, να πω δύο λόγια όσον αφορά το πλαίσιο ε, της ε, πρότασης που έκανα, ε, που ήταν πρόταση πρωτοβουλίας της Επιτροπής μας όσον αφορά την αποτελεσματικότητα και τη συνοχή της αναπτυξιακής βοήθειας και θα αναφέρω και κάποια ερωτήματα τα οποία μου φαίνονται σημαντικά στα πλαίσια της έκθεσης αυτής. Πρώτα απ' όλα, όπως άλλωστε το είπατε κι εσείς, στην προηγούμενη εντολή ήδη είχα την τιμή να είμαι ε, εισηγητής για το τέταρτο φόρουμ για την αποτελεσματικότητα της αναπτυξιακής ε, βοήθειας ε, που είχε σαν επιστέγασμα την εταιρική σχέση του Μπουζάν τότε είμαστε σε μία περίοδο σκέψης και θυμάμαι όλα τα, όλες τις συζητήσεις που κάναμε για το κατά πόσον σκόπιμο θα ήταν να περάσουμε από την γενικότερη έννοια της αποτελεσματικότητας στην πιο συγκεκριμένη έννοια της αποτελεσματικότητας της αναπτυξιακής βοήθειας. Και πέντε χρόνια μετά, το 2016, οι συζητήσεις αυτές έχουν εξελιχθεί και νομίζω ότι πλέον ε, έχουμε ενταχθεί στη λογική της ε, συνοχής της αναπτυξιακής ε, βοήθειας. Οι δεσμεύσεις του Μπουζάν προστιθέμενες και, προστιθέμενες και τις αποφάσεις της Άκρα και του Παρισιού μας έχουν οδηγήσει σε καλύτερη αντιμετώπιση της, της αποτελεσματικότητας οποιοδήποτε είδους βοήθειας. Ε, ε, η ιδιοποίηση και η ιδιοκτησία όπως λέμε των ε, αρχών από τις χώρες καθώς επίσης και η δυνατότητα επιλογών από πλευράς των είδων των χωρών το άνοιγμα των εταιρικών σχέσεων επί τη βάση της αμοιβαίας αξιοπιστίας οπωσδήποτε είναι ιδιαίτερα σημαντικά ακόμα σήμερα. Το Μπουζάν οπωσδήποτε αποτέλεσε ένα ποιοτικό άλμα ε, όσον αφορά τις ε, σχέσεις ε, των ε, χορηγών του ιδιωτικού τομέα, της κοινωνίας των πολιτών, όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως επίσης. Στο Μπουζάν είχαμε αναφερθεί ιδιαιτέρως στα ανθρώπινα δικαιώματα ε, και την ε, δημοκρατική ιδιοποίηση των αναπτυξιακών αρχών σε σχέση βεβαίως και με μια αποτελεσματική διοίκηση και την δημιουργία ενός μηχανισμού βάσει του οποίου θα μπορούσε να ε, προωθηθεί αυτή η συνεργασία και η συζήτηση, δηλαδή αναφέρομαι σε αυτήν την παγκόσμια συνεργασία για την ε, ε, αναπτυξιακή βοήθεια με τον τρόπο αυτό αλλάξαμε τον τρόπο σκέψης, αλλάξαμε το υπόδειγμα κατά κάποιο τρόπο, ε, περνώντας από μία ε, ε, αντιμετώπιση βορρά-νότου, δωρητών και απολαμβανόντων της βοήθειας, σε μία γενικότερη, συνολικότερη παγκόσμια αντιμετώπιση. Τώρα, στα πλαίσια της δεύτερης συνεργασίας υψηλού επίπεδου, που θα λάβει χώρα όπως υπενθυμίσατε και εσείς ε, κύριε Πρόεδρε τέλος του έτου στο Ναϊρόμπι ε, θεώρησα ότι είναι σημαντικό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ξαναδεί λίγο το θέμα όχι απλώς ε, γιατί θα πρέπει να υπάρξει μια συνέχεια στην αντιμετώπιση του θέματος, έστω και αν αντικειμενικά θεωρώ ότι θα πρέπει να δούμε οπωσδήποτε σε ποιο μέτρο ε, έχουν υλοποιηθεί οι δεσμεύσει του Μπουζάν, αλλά κυρίως γιατί ε, στα πλαίσια της υλοποίησης των, του, θεματολογίου της Αντίς Αμπέμπα και όσον αφορά δηλαδή και τη χρηματοδότηση της ε, βοήθειας, το θέμα της αποτελεσματικότητας της αναπτυξιακής σε ε, ε, παίρνει πολύ σημαντικές ε, διαστάσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί και παίζει ρόλο στην οικοδόμηση και θέσπιση των κριτηρίων αλλά και στα πλαίσια της, του θεματολογίου για το 2030 οφείλει να αναλάβει ηγετικό ρόλο όσον αφορά τα θέματα αυτά και όσον αφορά την συνέργεια μεταξύ των στοιχείων αυτών. Αυτό άλλωστε θα συζητηθεί ιδιαίτερος στο Ναϊρόμπι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάνει πολύ σημαντικά βήματα έτσι ώστε να ε, βελτιωθεί η διαφάνεια, ο προγραμματισμός, ε, το θέμα των ε, συγκρούσεων και των ευάλωτων χωρών, αλλά και όσον αφορά τα μετρήσιμα αποτελέσματα. Νομίζω ότι και εμείς οι ίδιοι θα πρέπει να το, να το αναγνωρίσουμε, γιατί μερικές φορές, και το έχω πει επανειλημμένα, μερικές φορές εμείς αυτομαστιγωνόμαστε. Ενώ έχουμε κάνει πολλά θετικά πράγματα και έχει υπάρξει πρόθεση τον Μάρτιο του 2015 ε, ε, ε, συμφωνήθηκαν οι αρχές και οι στόχοι για την αναπτυξιακή βοήθεια και βάσει αυτών η ορατότητα και η αποτελεσματικότητα της βοήθειας έχουν αυξηθεί. Βεβαίως θα πρέπει να αναλύσουμε ποια είναι τα στοιχεία τα οποία μπορούν να προωθηθούν ακόμα περισσότερα, αλλά παρόλα αυτά θα πρέπει να δούμε ότι οι βάσεις υπάρχουν υπάρχουν ε, και ότι οι βάσεις αυτές οδηγούν σε μια λογική τελείως διαφορετική από αυτή που είχαμε πέντε χρόνια πριν. Το έγγραφο προετοιμασίας ε, του Ναϊρόμπι ε, ακριβώς υπογραμμίζει την σημασία της παγκόσμιας εταιρικής σχέσης και θέτει τις βάσεις για το θεματολόγιο του 2030 όσον αφορά την συνολική συμμετοχή των χωρών και την επιτάχυνση. Γιατί αυτά τα δύο στοιχεία είναι πάρα πολύ σημαντικά. Εγώ θα ήθελα όμως κυρίως να αναφερθώ στη διασύνδεση και τις συνέργειες. Ο στόχος 17 των, ε, των βιώσιμων αναπτυξιακών στόχων καλεί ακριβώς τις κυβερνήσεις ε, για καλύτερη συνεργασία, κυρίως δε συνεργασία υπέρ ε, της αναπτυξιακής συνεργασίας. Ε, και ε, θα πρέπει να δούμε πώς ε, θα υλοποιηθεί αυτή η διασύνδεση. Υπάρχουν πολλές δυνατότητες μεταξύ των οποίων το παρατηρητήριο του Μπουζάν που θα πρέπει οπωσδήποτε να ενισχυθεί. Πιστεύουμε ότι και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στον Αϊρόμπι και στα πλαίσια της παγκόσμιας θετικής σχέσης θα πρέπει να ενταθούν οι προσπάθειες. Είμαι ευτυχής που έχω την ευκαιρία να κάνουμε τη συζήτηση αυτή και να ακούσω και την άποψη των συναδέλφων. Είναι πολύ σημαντικό να ακούσω τους ε, συναδέλφους γιατί βρισκόμαστε ακόμα στην αρχή της εργασίας. Ευχαριστώ πολύ ε, για τις παρεμβάσεις τους ε, και για τα όσα μας είπαν οι δύο κυρίες. Ναι βεβαίως βλέπω ότι πολλοί έχουν ζητήσει το λόγο από τους συναδέλφους. Όλοι αυτοί έχουν ζητήσει το λόγο. Θέλει να προσθεθεί κάποιο στον κατάλογο των αγορητών. Όχι, από ό,τι φαίνεται. Έχουμε χρόνο, λοιπόν. Ο Σέλβος Λίτς. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τους προβληματισμούς που κάνατε και τη δικασία του Μπουσάν και για το όσα προτείνετε για να προχωρήσουμε και για τις πολύ εξελιγμένες ιδέες σας, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει για τα πραγματικά νούμερα να τα πούμε έξω από τα δόντια. Θα ήθελα να δω καταρχήν τι υπάρχει σε επίπεδο κρατών μελών, τι μπορούμε να μάθουμε, από πού πρέπει να συνεχίσουμε και όπως είπατε και για την Ιταλία, να δούμε ποιες είναι οι βέλτιστες πρακτικές. Να δούμε δηλαδή σε ευρωπαϊκό επίπεδο τι μπορούμε να κάνουμε, να πιο συγκεκριμένη Τώρα, για την πρώτη δήλωση που κάνατε. Θα ήθελα να σχολιάσω τα όσα είπατε για τον ιδιωτικό κλάδο που έχει και αυτός ένα σημαντικό ρόλο που πρέπει να αναλάβει. Συμφωνώ μεν πως ο ιδιωτικός κλάδος πρέπει να κάνει παραπάνω, αλλά είπατε πως η χρηματοδότηση ε, στο σημείο αυτό μέσω πρωτοκόλλων θα πρέπει να ενισχυθεί. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό για σας, πώς μπορούμε εμείς να περιγράψουμε ποια είναι αυτά τα χρηματοδοτικά εργαλεία και πώς μπορούμε να τα προκοδοτήσουμε περισσότερο, πώς μπορούμε να γνωρίζουμε εμείς ποιοι είναι οι οικονομικοί στόχοι αυτών των χωρών, τι σημαίνει για το πακέτο, για το ε, κλίμα ένα τέτοιου είδους, ε, μια στόχευση. Τι σημαίνει για τις ε, γυναίκες, ε, τι σημαίνει ε, για την οικονομική διακυβέρνηση. Καλό είναι να τα περιγράφετε, αλλά θα πρέπει να έρθετε και σε επαφή με τις χώρες εταίρους για να δούμε ποιοι είναι οι δικοί τους στόχοι και ποιες είναι οι οικονομικές ανάγκες που προκύπτουν από τους στόχους αυτούς. Και για να μιλήσω για το θέμα Concord, να δούμε ποιοι είναι οι μηχανισμοί επιτήρησης και χρηματοδότησης οι οποίοι μπορούν βήμα-βήμα να μας φέρουν σε ε, απτά αποτελέσματα. Σας ευχαριστώ λοιπόν για όλες αυτές τις ε, ε, δηλώσεις και κύριε Πρέντε σας ευχαριστώ που είστε τόσο ανοιχτός ίσως θα έπρεπε να κάνουμε κάποιο brainstorming έτσι ώστε οι συνάδελφοι να μπορέσουν να τονίσουν τα σημεία αυτά ξέρετε πως είναι κρίσιμα είναι μια πολύ καλή ευκαιρία πριν το Ναϊρόμπι να γίνουν κάποια θέματα πιο ορατά και να δείξουμε πως η Ευρώπη θέλει να κάνει πραγματικά βήματα πιο συγκεκριμένα Σας ευχαριστώ Ευχαριστώ πολύ η κυρία Θεοχάρους I will speak in Greek, so please put your headphones on. Ε, θα ήθελα να πάω λίγο πιο πέρα από το πνεύμα της έκθεσης και την τεχνοκρατική αντίληψη που επικρατεί συνήθως. Is it okay? Shall I start from uh, Θα ήθελα να πάω λίγο πιο πέρα από, την, από το πνεύμα της έκθεσης και την τεχνοκρατική αντίληψη που επικρατεί ε, συνήθως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ειδικότερα στην Επιτροπή μας. Να ευχαριστήσω και τις δυο σας για την συζητήσεις. Θέλω να σας πω ότι ήμουνα και στο Μπουζάν και εκεί είχα εκφράσει τις ίδιες ανησυχίες που θα πω και σήμερα και υπήρξα και εκπρόσωπος αρκετών NGO στην Concord και ίσως να είμαι ακόμη δεν το ξέρω αν είμαι ε, κάπου καταγεγραμμένη. Ε, θα επιμείνω ότι η έλλειψη αποτελεσματικότητας οφείλεται στην άγνοια των πραγματικοτήτων στο πεδίο και σε κάθε περιοχή ξεχωριστά. Δεν τίθενται προτεραιότητες για την επιτέλεση ε, την διάθεση της αναπτυξιακής ε, βοήθειας. Για παράδειγμα, όταν αύριο θα είμαστε στο Ναϊρόμπι, εγώ θα ήθελα αντί να κλειστούμε μέσα στο Hilton ή στο Convention Center που θα μας έχουν, να πάμε μια βόλτα στα slum cities γύρω-γύρω από το Ναϊρόμπι για να δείτε ποια είναι πραγματικότητα. Ότι για να αντιμετωπίσεις τη γαστρεντερίτιδα δεν μπορεί να δίνεις βαϊόφιλους, συνεχώς, αλλά πρέπει να τους σταματήσεις από το να παίρνουν νερό από τα αυλάκια, από τα κανάλια και να, να το πίνουν, γιατί τα αυλάκια τους είναι switch systems και εκεί μέσα καταλήγουν όλα τα, όλα τα απόβλητα των slum cities. Ε, επίσης, αυτό που λέμε ότι πρέπει να έχουν λόγο οι πολίτες και η κοινωνία των πολιτών. Αν ρωτήσετε τον οποιοδήποτε γιατρό σε ένα μικρό νοσοκομείο της Αφρικής τι είναι εκείνο που θέλει να του δώσετε, θα απαντήσει αμέσως λαπαροσκόπικ system. Θέλουν όλοι να κάνουν λαπαροσκοπικές επεμβάσεις τη στιγμή που δεν έχουν νηστέρια να κάνουν τις κλασικές επεμβάσεις. Καταλαβαίνετε ότι εμείς πρέπει να θέσουμε και κάποιες προτεραιότητες στη βάση της γνώσης και της εμπειρίας που υπάρχει μέχρι τώρα. Όσον αφορά τις κυβερνήσεις, συνεχώς προβάλλουν νομικούς φραγμούς, Εδώθησαν φέτος 10 projects των 20 εκατομμυρίων το καθένα σε 10 αφρικανικές χώρες, σε όλες τις αφρικανικές χώρες, αλλά 10 θα μπορούσαν να τα διεκδικήσουν. Λίγη προθεσμία σήμερα για φωτοβολταϊκά συστήματα μετατροπής της ηλιακής ενέργειας, όχι σε ηλεκτρική που σταματάει με το που πέφτει ο ήλιος, αλλά σε θερμική που συνεχίζει να δουλεύει και όλη τη διάρκεια της νύχτας. Καμία χώρα δεν κατάφερε να το πάρει και ακόμη και η Ρουάντα στην οποία είχα προσωπική εμπλοκή και τους είχα συγγράψει ακόμη και την αίτηση έληξε η προθεσμία και μου είπαν ότι το νομικό πλαίσιο δεν τους επιτρέπει να κινηθούν προς αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή όταν δεν υπάρξουν ε, ε, reforms προς την κατεύθυνση της, ε, της βελτίωσης της νομολογίας κάθε χώρας για να μπορεί να αποδέχεται τη βοήθεια Καταλαβαίνετε ότι δεν πρόκειται να πάμε πουθενά δημιουργώντας έργα υποδομής που θα σταματήσουν την υποανάπτυξη και θα δώσουν ε, ε πραγματική όθηση στην ε, πρόοδο ε, της, κάθε περιοχής. Υπάρχει μια μικρή περίπτωση να προλάβει η Αίγυπτο σήμερα και να πάρει η Αίγυπτος αυτό το σύστημα το μοναδικό από τα 10 που, που, που θα δοθεί στην Αφρική. Βεβαίως η Αίγυπτος δεν ανήκει στις χώρες που συνήθως μας απασχολούν. Ε, οι χώρες αυτές επιδίδονται κυρίως σε έργα βιτρίνας και η αναπτυξιακή βοήθεια πολλές φορές όταν διοχετεύεται μέσα από τις κεντρικές κυβερνήσεις εάν δεν γίνεται, εάν δεν πέφτει θύμα της διαφθοράς που συνήθως επικρατεί θα μετατραπεί σε έργα βιτρίνας. Είναι γι' αυτό που επιμένω ότι πρέπει να κινούμαστε προς τις μικρές κοινότητες, προς την περιφέρεια προς τις τοπικές αρχές σε επίπεδο δημιουργίας συγκεκριμένων ε, έργων υποδομής. Ε, βεβαίως πιστεύω ότι ε, έχει γίνει σημαντική πρόοδος, δεν μπορώ να τα μηδενίσω όλα. Για παράδειγμα, όσον αφορά το AIDS, την παιδική θνησιμότητα, την περιγεννητική θνησιμότητα, τη θνησιμότητα των γυναικών κατά τη διάρκεια του τοκετού, έχει υπάρξει ε, βελτίωση. Οι εμβολιασμοί έχουν καλύψει σημαντικό, ε, σημαντικό επίπεδο, αλλά όταν για παράδειγμα ένας ασθενής που για να πάρει τα φάρμακα του AIDS δωρεάν πρέπει να διανύσει μία απόσταση 6 ώρων με τα πόδια για να φτάσει στη στάση του λεωφορείου που θα τον πάρει άλλες 6 ώρες και να κάνει ανάλυση αν όντως έχει AIDS, ότι είναι HIV positive για να του δώσουν τα φάρμακα, γιατί ξέρετε ότι η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας δεν τα δίνει τα φάρμακα αν δεν υπάρχει αυτή η απόδειξη. Ε, η, η, η εργαστηριακή επιβεβαίωση είναι σίγουρο ότι αυτός ο άνθρωπος δεν θα φτάσει ποτέ στο σημείο να πάρει τα φάρμακα. Δίνουμε τα φάρμακα, αλλά σε ποιου, χωρίς να υπάρχει η απαραίτητη υποδομή. Είναι η υποχρέωση μας να χρησιμοποιήσουμε τεχνοκράτες και ανθρώπους που γνωρίζουν την κάθε μια περιοχή και να μην λέμε ότι δίνουμε ένα τεράστιο ποσό είτε από ιδιωτικού τομεί, είτε από φιλανθρωπικού αφάντ, ε, είτε από ε, την Ευρωπαϊκή Ένωση και έτσι έχουμε καλύψει τη συνείδησή μας ότι κάναμε το καθήκον μας σωστά. Είναι εκείνο που έχει πιο μεγάλη σημασία είναι να επενδύσουμε στην εκπαίδευση τους και στην βελτίωση της υγείας τους, αλλά με την δική μας παρουσία εκεί πέρα των τεχνοκρατών μας και του Task Force, το οποίο θα πρέπει να είναι παρόν και να διοχετεύει τη βοήθεια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Σαρ Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Αυτή η συζήτηση καταδεικνύει ότι η αποτελεσματικότητα της ανθρωπιστικής βοήθειας είναι και τεχνικό αλλά και ιδιαίτερα πολιτικό θέμα. Αυτά που μας απασχόλησαν σήμερα σε μεγάλο βαθμό ε, είναι τεχνικού χαρακτήρα αυτός ο συνδυασμός, περισσότερη αποτελεσματικότητα και να ε, επιδιώκουμε αποτελέσματα. Θεωρώ ότι σε αυτά τα τεχνικά θέματα έχει υπάρξει ουσιώδης πρόοδο και ο σίγουρα ε, πρέπει να επενεθεί γιατί ξεκίνησε αυτή τη διαδικασία. Είναι ο πρώτος ε, μεγάλης κλίμακας διεθνής οργανισμός που ήδη από τη δεκαετία του 1990 έπαιξε πρωτοπόρο ρόλο στην ε, διαδικασία αποτίμησης των αναπτυξιακών πολιτικών. Αλλά αυτό είναι θέμα αποτελεσματικότητας. Είναι ένα στοιχείο της μεθόδου ΩΣΑ για να μετρήσουμε την αναπτυξιακή βοήθεια. Έχουμε λοιπόν το πόσο κατάλληλη είναι η αποτελεσματικότητα, το μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα και η βιωσιμότητα. Κυρίως συζητάμε την βράχη πρόθεσμη αποτελεσματικότητα, δηλαδή καλύτερο αποτέλεσμα με λιγότερους πόρους, καλύτερο αποτέλεσμα με πιο απλές διαδικασίες, ιδιαίτερα όσον αφορά το συνδυασμό των δικών μας ε, στόχων με τους στόχους της χώρας και για να αποφεύγουμε την επικάλυψη. Αλλά για να είμαστε πραγματικά μακροπρόθεσμα αποτελεσματικοί πρέπει να κάνουμε περισσότερα. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι χώρες ε, που λαμβάνουν τη βοήθεια και ο ΩΣΑ, όλοι μας, είμαστε και τμήμα του προβλήματος και τμήμα της λύσης. Της λύσης είπα πώς. Ο ΩΣΑ νομίζω έκανε ό,τι μπορούσε για να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα. Αλλά η μακροπρόθεσμη αποτελεσματικότητα πρέπει να γίνει με βάση ε, μια ευρύτερη αντιμετώπιση του ρόλου, του ρόλου και αυτών που δίνουν βοήθεια και αυτών που λαμβάνουν βοήθεια. Ε, η μεγάλη πρόκληση για το άμεσο μέλλον είναι η μείωση των ανισοτήτων. Και πώς μπορούν να μειωθούν οι ανισότητες είναι να βελτιωθεί ε, ο τρόπος συλλογής φορολογικών πόρων από τη μία μεριά και από την άλλη μεριά η πρόσβαση στις ε, κοινωνικές υπηρεσίες. Για να γίνουν περισσότερα εδώ πρέπει όλοι να κατανοούμε με τον ίδιο τρόπο το πρόβλημα. Και εδώ είναι το θέμα. Ορισμένοι θεωρούν ε, ότι το θέμα της πρόσβασης στις κοινωνικές υπηρεσίες πρέπει να αντιμετωπιστεί με τον Α, άλλοι με τον Β τρόπο. Για παράδειγμα, στι ΗΠΑ ορισμένοι αμφισβητούν ακόμη και την ε, ε, περιορισμένη πρόοδο που έχει επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια όσον αφορά την πρόσβαση στις κοινωνικές υπηρεσίες. Πρέπει πραγματικά να πιέσουμε το G20 γιατί τα μέλη του G20 ε, που δεν καταφέρνουν να συμφωνήσουν είναι και μέλη του ΟΣΑ. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει περισσότερη σύγκληση απόψεων στα πλαίσια του ΟΣΑ και στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με κάθε σεβασμό ε, και σας ευχαριστώ για τη σταυμάσια παρουσία σας και, και τις δύο σας ευχαριστώ αλλά πρέπει να δούμε ευρύτερα το θέμα δεν είναι μόνο μεθοδολογικά τα προβλήματα, δεν είναι μόνο τεχνικής φύσης, δεν είναι μόνο ε, διαδικαστικά. Πρέπει να γίνουν ε, ευρύτερα πολιτικές συζητήσεις που δεν είναι εύκολο, αλλά επειδή δεν είναι εύκολο δεν σημαίνει πως πρέπει να το αγνοήσουμε. Ευχαριστώ η Λόλα Σάντσε. Ευχαριστώ, Λίντα. Είναι 10 χρόνια που ορισμένες αντισώμενες χώρες και οι αναπτυγμένες χώρες ε, υπέγραψαν τη διακήρυξη των Παρισίων αποτελεσματικότητα. Όπως είπε ο κύριο Πρέντα, ορισμένα πράγματα έγιναν καλά, αλλά τώρα πρέπει κυρίως να ασχοληθούμε με τις αδυναμίες και να βελτιώσουμε την κατάσταση. Όλες τις φάσεις της ε, χορήγησης ε, της βοήθειας είναι δύσκολο να δούμε σε τι βαθμό επιτύχαμε τους στόχους. Μια έκθεση του 2014 λέει ότι δεν μπορούμε να διαπιστώσουμε κατά πόσο έχουμε σημειώσει πρόοδο, γιατί μας λείπει επαρκής πληροφόρηση. Και τα λίγα στοιχεία που έχουμε λένε ότι μόνο μερικά έχουμε επιτύχει τις δεσμεύσεις μας. Ιδιαίτερα οι χώρες χορηγοί. Αυτό οφείλεται σε διάφορες ε, αιτίες. Πρώτα απ' όλα όλο και περισσότερο ε, ασχολούμεθα λιγότερο με τα θέματα. Έχει υπάρξει βέβαια αλλαγή ε, εστίασης μετά τον Μπουζάν. Αλλά επειδή τον Μπουζάν ε, έβαλε περισσότερους στόχους, τελικά ασχολούμεθα λιγότερο με τον καθένα. Πρέπει λοιπόν όμως ό,τι έχουμε αποφασίσει να εκπληρώσουμε, να το κάνουμε. Και ακόμη και οι χώρες χορηγοί. Διαπιστώνουμε ότι μειώνεται ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από την συνάντηση των Μπουζάν τότε στη συνάντηση στο Μπουζάν η Ευρωπαϊκή Ένωση έπαιζε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έπαιζε συγκεκριμένο ρόλο και στα πλαίσια της Επιτροπής Ανάπτυξης του ΟΣΑ αλλά μέσω, της, μέσω δηλαδή της αγωγής συγκεκριμένων προτάσεων. Παράδειγμα, είχαμε την Ευρωπαϊκή Συνένεση για την Ανάπτυξη, αλλά τα τελευταία χρόνια δεν ε, παίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτό το ρόλο συντονισμού και καμία χώρα δεν έχει αναλάβει να παίξει αυτό το ρόλο. Χρειάζεται επίσης να υπάρχει περισσότερη ενασχόληση με την ουσία. Ο κύριος Μαλέκ, ε, που είναι υπεύθυνο της ομάδας για την ε, αποτελεσματικότητα της βοήθειας είπε ότι πρέπει να αλλάξει η συμπεριφορά. Πρέπει να υπάρχει περισσότερη προετοιμασία για τη λήψη βοήθειας. Οι περισσότεροι χορηγοί δεν ε, έκαναν ουσιώδεις αλλαγές, μόνο διακοσμητικές. Επιπλέον, ο τρόπος χορήγησης βοήθειάς μας έχει αλλάξει. Δεν δίνουμε απευθείας βοήθεια στον προϋπολογισμό των χωρών. Απλώς μιλάμε περισσότερο για συνεργασία τη χρηματοδότηση. Αυτό το περίφημο blending, όπου συμμετέχει και ο ιδιωτικός ε, τομέας, που δεν είναι τόσο αποτελεσματική αυτή η μέθοδος. Και δεν ξέρουμε και πού πάμε. Είναι περιορισμένη η γνώση που έχουμε για το κατά πόσο επιτυγχάνουμε. Χάνουμε στην ουσία αποτελεσματικότητα ασχολούμεθα περισσότερο με τους στόχους της ε, βιώσιμης ανάπτυξης και κυρίως ασχολούμεθα με την κλιματική αλλαγή και πολλοί έχουν μια ειδοληψία με τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα. Υπάρχουν πολλές αμφιβολίες. Τώρα έχουμε την ε, προσπάθεια ε, καθορισμού των στόχων του 2030. Άρα η αποτελεσματικότητα πρέπει να παίξει μεγαλύτερο ρόλο να μην ξεχάσουμε ποιε είναι οι βασικέ αρχέ που συμφωνήσαμε στο Παρίσι. Υπάρχει ανάγκη να βελτιώσουμε την επίπτωση της βοήθειας στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων. Κύριε Ισηγητά, σας παρακαλώ να λάβετε υπόψη αυτές τις ανησυχίες και ελπίζω στην Επιτροπή μας να κάνουμε ό,τι μπορούμε, ούτω ώστε να επιτύχει το και όλε αυτέ οι φιλόδοξε διακηρύξεις να έχουν συγκεκριμένη μετάφραση σε δράση με σαφή στόχο κάθε χορήγηση βοήθειας για την ανάπτυξη πρέπει να σέβεται τις αρχές της αποτελεσματικότητας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ η Χάιντι Χάουταλα. <clears throat> Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και εγώ ήμουν στον Μπουζάν. Ήμουν υπουργό ε, στην κυβέρνηση της Φιλανδίας για την ε, διεθνή ανάπτυξη. Και θυμάμαι ότι ένα από τα κύρια σημεία τριβή ήταν πώς να καταλάβουμε και πώς να αναγνωρίσουμε τον ουσιώδη ρόλο της κοινωνίας των πολιτών. Αυτό πρέπει να μας απασχολήσει περισσότερο και να αποφασίσουμε να τον ενισχύσουμε στον αερόμπι. <clears throat> Επίσης υπάρχουν προκλήσεις τώρα για τις χώρες BRICS και πολλές άλλες χώρες του Νότου. Και ίσως για πολλές από αυτές τις χώρες η ε, αντίληψη που έχουν για τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών να είναι διαφορετική από τη δική μας. Άρα θα πρέπει να συνεχίσουμε να προωθούμε το θέμα αυτό. Ήταν θετικό στον Μπουζάν ότι η Ινδία και η Κίνα, αν θυμάμαι καλά, συνέβαλαν στην ε, διαμόρφωση των πορισμάτων και προσυπέγραψαν τελικά. Θα ήθελα να μας πούν οι ομιλητές μας Με ποιο τρόπο η συμμετοχή τέτοιων χωρών BRICS άλλαξε συνολικά το πλαίσιο της αναπτυξιακής συνεργασίας. Γιατί πρέπει οπωσδήποτε να ενταχθούν και αυτές οι χώρες σε αυτό το πλαίσιο. Αλλά ορισμένες φορές έχουν εντελώς διαφορετικές προτεραιότητες. Εντελώς διαφορετικές αρχές. Κάτι άλλο της διαδικασίας αυτής που οδηγεί από τον Μπουζάν στον Αερόμπι είναι πώς έχουν εφαρμοστεί τα, οι λεγόμενες δομικές μονάδες του Μπουζάν. Μπουζάν Building Blocks. Να αναφέρω μερικές που θεωρώ σημαντικές. Για παράδειγμα, τα ε, κράτη που κινδυνεύουν να καταρρεύσουν, fragile states, τι κάναμε για να τα βοηθήσουμε. Κάτι άλλο σημαντικό, που δεν νομίζω ότι έχει αναφερθεί ακόμη τη συζήτηση στο κοινοβούλιο μας είναι να μειωθεί ο κατακαιρματισμός της αναπτυξιακής βοήθειας. Δίνουμε πολλά λεφτά, αλλά πολλές φορές ε, δίνονται υπερβολικά πολλούς ε, λήπτες. Έχει υπάρξει μείωση του κατακαιρματισμού της βοήθειας. Αυτή είναι η ερώτησή μου. Και κάτι άλλο που είναι πραγματικά ιδιαίτερα σημαντικό. Πρέπει η προσέγγιση μας να βασίζεται σε δικαιώματα. Δεν ήταν προφανές αυτό στη συζητήση των Μπουζάν, λόγω της ευρύτητας των συμμετεχόντων. Θεωρώ ότι αυτή η παγκόσμια εταιρική σχέση για την συνεργασία, για την ανάπτυξη, για την αποτελεσματικότητα της συνεργασίας, για την ανάπτυξη είναι σημαντική και οι αρχές των Παρισίων, της Ακρά και του Μπουζάν πρέπει να εφαρμοστούν. Σας ευχαριστώ που μας εξηγήσατε τις αδυναμίες στην εφαρμογή. Πρέπει να μας απασχολεί μονίμως αυτό το θέμα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ η Μαρία Χόιμπουκ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για την ε, πλούσια πληροφόρηση που μας δώσατε. Η Χάιντι Χάουταλα αναφέρθηκε στον κατακαιρματισμό δίνουμε λεφτά προς πάρα πολλές κατευθύνσεις. Σωστό, συμφωνώ. Κάτι που με ανησυχεί ιδιαίτερα είναι η συζήτηση για τη μετανάστευση που οδηγεί ότι δεν ασχολούμεθα πια με αυτές τις αρχές της αποτελεσματικότητας. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αγνοούμε εντελώς σταδιακά. Λαμβάνονται πολλά μέτρα για την αποφυγή της μετανάστευσης και χρησιμοποιώ αυτό τον όρο. Αποφυγή, όχι διαχείριση της μετανάστευσης. Όλα αυτά δίνονται μέσω ειδικών ταμείων που είναι εκτός ε, του ενωσιακού προπολογισμού και δεν υπάγονται στον κοινοβουλευτικό μας έλεγχο. Και αυτό είναι μόνο ένα θέμα. Άρα πέρα από την αρχή της αποτελεσματικότητας και την ανάγκη ε, αμοιβαίας λογοδοσίας πώς μπορούμε να θεωρήσουμε ότι συνδυάζονται με τους στόχους των χωρών και γίνονται αποδεκτά από τον πληθυσμό τα μέτρα αυτά. Γενικότερα, η συνολική στρατηγική που υποβλήθηκε τον ε, Ιούνιο από το Αναπτυξιακό Ταμείο περιλαμβάνει και παραθέτω ότι πρέπει να είναι πιο ελαστική και η μακροχρόνη κύκλοι προγραμματισμού Πρέπει να γίνουν πιο ευέλικτοι και πρέπει να αξιοποιούμε περισσότερο ειδικά ταμεία. Σήμερα το πρωί ακούσαμε τον Κούντουνς ότι ο μακροπρόθεσμος χαρακτήρας και η αξιοπιστία της χρηματοδότησης είναι πολύ θετικά στοιχεία. Και τώρα θέλουμε περισσότερη ελαστικοποίηση. Πώς συνδυάζονται αυτά τα δύο. Είναι ισότιμη αυτή η συνεργασία. Όταν εμείς ε, ταχύτατα και ανάλογα με τα παροδικά συμφέροντα κάποιων χωρών ανοίγουν ή κλείνουν τις στρόφιγγα της χρηματοδότησης. Έχω ανησυχίες γι' αυτό. Και παρακαλώ τον εισηγητή να περιλάβει στην έκθεσή του και αυτά τα θέματα και να ασχοληθούμε με τις παρούσες παγκόσμιες προκλήσεις. Για να έχουμε ουσιώδες πρόγραμμα για το 2030 χρειάζεται παγκόσμια συνεργασία και μάλιστα περισσότερη, όχι λιγότερη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Έχουμε ε, την ε, εκπρόσωπο της ΔΙΖΙΝΤΕΦΚΟ υπεύθυνη για την αποτελεσματικότητα της ανθρωπιστικής βοήθειας, ε, Σαντάλ. ναι, ναι, η ομάδα μου προετοιμάζεται για τον Ναϊρόμπι τώρα. θα ήθελα να σας δώσω μια επικαιροποιημένη ιδέα για το πού βρισκόμαστε, τι κάνουμε στις προετοιμασίες μας για το Ναϊρόμπι. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι μέλος της Steering Committee του GPDC. Έχουμε έχουμε τρεις συνπροέδρους, ε, σύντομα θα γίνουν τέσσερις οι συμπροέδροι, γιατί η Steering Committee αποφάσισε να έχει και έναν τέταρτο. civil society, parliamentarians, ε, έτσι ώστε να έχουμε και εκπρόσωπο των τροπικών οργανώσεων. Οπωσδήποτε θα προετοιμαστούμε μαζί με το Συμβούλιο και βεβαίως ε, ε καλωσορίζουμε και την έκθεση του κυρίου Πρέντα εξ ονόματος ε, του ε, Κοινοβουλίου εν ώψη του Ναϊρόμπι. Έχουμε και ένα άλλο έγγραφο το οποίο έχει εκπονήσει ο ε, πρέσβης Κεμάλ εξ ονόματος ε, της διοργανώτριας ε, Κένιας και εκεί αναφέρονται κάποια, κάποιοι ιδιαίτερα φιλόδοξοι στόχοι όπου η παγκόσμια εταιρική σχέση εγγράφεται ως κύριο συστατικό των, του, του θεματολογίου για το 2030. Πιστεύουμε ότι το παράδειγμα το οποίο έχει δοθεί από την ανθρωπιστική διάσκεψη, ανθρωπιστική διάσκεψη ε, κορυφής ε, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ως ένας καλός τρόπος ε, για να προχωρήσουμε. Ε, βεβαίως τα στοιχεία τα ανθρωπιστικά είναι ιδιαίτερος παρόντα στη συνολική εταιρική σκέψη, αλλά βεβαίως θα πρέπει να ενταχθεί περισσότερο και ο ιδιωτικό τομέα, αλλά και οι αναδυόμενες οικονομίες, ε, οι χώρες μέσου εισοδήματος, έτσι ώστε να ε, κατανοήσουμε καλύτερα το περιβάλλον στο οποίο ε, κινούνται ε, όλοι αυτοί οι πρωταγωνιστές και επομένως θα πρέπει να συνεμπλακούν στην διαδικασία. Επίσης χρειαζόμαστε μια ολοκληρωμένη διαδικασία η οποία δεν θα βασίζεται μονάχα στη Νέα Υόρκη αλλά θα λαμβάνει υπόψη και άλλες τις, τις άλλες γεωγραφικές ε, περιοχές ε, οι οποίες εμπλέκονται. Πολλά λοιπόν θα πρέπει να γίνουν ακόμα ε, όσον αφορά το τελικό έγγραφο, μια επόμενη εκδοχή του οποίου αναμένουμε για τα μέσα Σεπτεμβρίου και βεβαίως θα υποβληθούν και θα υποβληθεί και σε εσά έτσι ώστε και θα σας ακοινοποιηθεί Η Προεδρία θα προετοιμάσει και τα συμπεράσματα του ε, ε, Συμβουλίου ε, σε σχέση με το HLM και βεβαίως δουλεύουμε σε συντονισμό με τα κράτη-μέλη και στα πλαίσια ενός τεχνικού σεμιναρίου που θα οργανωθεί ε, περί τα τέλη Σεπτεμβρίου, 21 Σεπτεμβρίου συγκεκριμένα, ε, έτσι ώστε να συνυπολογιστούν και συνεκτιμηθούν όλα τα στοιχεία. επίση. θα υπάρξει μια άλλη έκθεση για να δούμε ε, πού ακριβώ βρισκόμαστε σαν Κομισιόν και σαν κράτη-μέλη όσον αφορά την υλοποίηση των δεσμεύσεων που έχουμε λάβει. Το ίδιο κάναμε και 24 μήνες πριν, όσο πλησιάζει το Ναϊρόμπι θα ενισχυθεί η διαδικασία αυτή για να ξέρουμε ακριβώς πού βρισκόμαστε. Υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα το οποίο είναι πολύ σημαντικό στην τελική ευθεία για τον Αϊρόμπι αλλά θα παίξει σημαντικό ρόλο και μετά τον Αϊρόμπι. Η εντολή ε, τη της συνολικής εταιρική ε, σχέσης ε, γιατί θα είναι κατά κάποιο τρόπο η διασύνδεση με το θεματολόγιο για το 2030. Χρειαζόμαστε μεγαλύτερη εστίαση στην υλοποίηση αναχώρα. Θέλουμε να είμαστε βέβαιοι ότι η επιτήρηση, το monitoring ε, θα είναι σωστό, η διασύνδεση με το θεματολόγιο του 2030 ε, και το follow-up θα ε, είναι σωστά και θα είναι ιδιαίτερο συνδεδεμένα με τις υποχρεώσεις λογοδοσίας του θεματολογίου του 2030. Οι συζητήσεις θα αφορούν το πεδίο εφαρμογής, τη συμπληρωματικότητα ε, και την εντολή για την συνολική εταιρική σκέψη. Αναφέρθηκα ήδη στην έκθεση την οποία θα εκπονήσουμε αλλά να σας πω επίσης ότι προετοιμαζόμαστε ε, και για την, ε, ε, και για την συνεδρίαση για το HLM, το οποίο συνδέεται άμεσα με το θεματολόγιο 2030 και στα πλαίσια αυτά και, να σας πω επίσης ότι εμπλεκόμαστε και με σειρά άλλων ε, πρωτοβουλειών που συνδέονται με αυτά τα building blocks του Μπουζάν που αναφέρθηκαν ε, προηγουμένως. Ε, έχουμε κοινέ συμπράξεις, έχουμε επίσης και την, μια πρόσφατη διάσκεψη σχετικά με την ενίσχυση και επιτάχυνση των κοινών συμπράξεων, έτσι ώστε και να σας πω ότι οι κοινέ δράσεις θα αποτελέσουν ε, τμήμα της ε, νέας ε, συνένεσης του τρόπου δηλαδή με τον οποίο συνεργαζόμαστε. Αυτά σύντομα για να σας πω που ακριβώς βρισκόμαστε. Έχουν υποβληθεί πολλές ερωτήσεις. Α, κύριε Γκέρεν, θέλετε κάτι άλλο. Ναι, μία ερώτηση σχετικά με την απουσία της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης από την σημερινή συνεδρίαση. μπορεί να συμβεί βέβαια αλλά μπορούμε να ε, ε, θεωρήσουμε ότι ε, όλες οι, όλες οι απόψεις που εκφράστηκαν από την Κομισιόν ταυτίζονται με τις απόψεις της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης Κομισιόν, ναι, όσον αφορά την συνεργασία και την αποτελεσματικότητα της συνεργασίας, κυρίως δε όσον αφορά τον κοινό προγραμματισμό που γίνεται ακριβώς από κοινού, έχουμε ταύτιση απόψεων με την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και επομένως δεν πρέπει να ανησυχείτε. Η κυρία Μπόσα πρώτα θα πάρει το λόγο και μετά ε, θα δώσω το λόγο στην επόμενη ομιλία της κυρίας Λεγουά. Ευχαριστώ πολύ. Ε, πολλά σχόλια, πολλές ε, περισσότερο από ερωτήσεις. Ε, με μεγάλη ευχαρίστηση ακούσαμε όλα αυτά τα στοιχεία και τα στοιχεία τα οποία μας είπε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όσον αφορά ορισμένα από τα θέματα που έθιξε ο κύριος Λίτς, ο οποίος δυστυχώς δεν είναι εδώ, πρέπει να σας πω ότι ναι, όντως εμείς θέλουμε να είμαστε πιο σαφείς και πιο απτοί όσον αφορά την αποτελεσματικότητα και τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να επιτύχουμε περισσότερα αποτελέσματα. Ε, ε, και ένας άλλος συνάδελφος είπε ότι δεν γίνονται αρκετά και δεν είναι ορατά. Όχι, εγώ πρέπει να σας πω ότι στην ουσία αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να επιτηρούμε όλες τις ε, περιοχές στις οποίες μπορούν να υπάρξουν διακυβεύματα. Ήδη στην έκθεση του 2014 αναφέραμε την, τις περιοχές αυτές, τα στοιχεία αυτά, τα οποία αποτελούσαν σημεία πρόθεσης και στην έκθεση του 2016 επίσης θα αναφέρουμε κάτι τέτοιο. Ε, και η Σούζαν το είπε προηγουμένως. Έχουμε αυτή την πλατφόρμα όπου αναφέρονται και περιλαμβάνονται όλα αυτά τα ε, στοιχεία και που αναφέρουμε βεβαίως και τις ε, επικρίσεις μας στις περιοχές οι οποίες δεν έχουν προωθηθεί καλά. Πρέπει να δείτε τις εκθέσεις αυτές έτσι, έτσι ώστε να έχετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες είναι γεγονός ότι εδώ πρόκειται και για μια πολιτική ατζέντα και επομένω έχει υπάρξει ένα είδος διήθηση, ας πούμε του ε, ε, λεξιλογίου αλλά ε, παρόλα αυτά στα συμπεράσματα της έκθεσης ε, οι αναφορέ είναι σαφείς. Σε σχέση και με αυτό που είπε η Σούζαν δεν είναι τόσο, κακό, δεν είναι τόσο κακή η γενική εικόνα. Εγώ δεν θέλω εδώ να περιγράψω με ιδιαίτερα θετικά χρώματα την όλη κατάσταση αλλά παρόλα αυτά ε, νομίζω εάν δείτε λίγο ε, την κατάσταση ε, θα δείτε ότι πραγματικά όλες οι, όλες οι αναπτυξιακές συνεργασίες βασίζονται σε πολλά θετικά στοιχεία. Έχει αλλάξει ο τρόπος διατύπωσης, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχει υπάρξει σημαντική πρόοδος. Αυτό δεν σημαίνει ότι εάν δεν έχουμε επιτύχει 100% τους στόχους, δεν έχουμε κάνει, δεν, έχουμε, δεν έχει υπάρξει βελτίωση βελτίωση όσον αφορά πολλούς πολλές παραμέτρους και πολλούς ε, δείκτες. Είναι αλήθεια ότι ε, υπάρχει μία τελμάτωση σε αυτή την ε, περίοδο, αλλά όταν μιλάμε για προβλεψιμότητα της αναπτυξιακής βοήθειας, αν υπάρχουν χώρες οι οποίες δεν θέλουν να δώσουν στοιχεία όσον αφορά την ευθυγράμμισή τους, σημαίνει, αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να μην υπάρχει απλή δέσμευση, αλλά να προχωρήσουμε προχωρήσουμε και σε κάποιες ε, ε, δομικές ε, αλλαγές. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Χρειαζόμαστε αυτό το ποιοτικό άλμα ε, πρέπει να περιγράψουμε ε, τα διακυβεύματα, πρέπει να δούμε ποιες είναι οι δομικές αυτές μεταρρυθμίσεις οι οποίες ε, μπορούν και πρέπει να οδηγήσουν σε νέες δεσμεύσεις. Είπατε ότι υπάρχει μια τεχνική, ένα τεχνικό θεματολόγιο με πολιτική διάσταση. Ναι, και επομένως είναι γεγονός ότι θα πρέπει να συμπεριληφθούν και θεωρήσεις όσον αφορά ε, το φορολογικό σύστημα, όσον αφορά το ασφαλιστικό σύστημα κτλ. Ε ε, ε, ε, πρέπει να σας πω ότι, ε, και, ε, ότι το, το θέμα της ε, εσωτερικής φορολογικής δομής και των ιδίων πόρων, των εγχωρίων πόρων, αποτελεί πλέον από τα πρώτα στοιχεία για, την, για το θεματολόγιο της ανάπτυξης. Κοιτάξτε, δεν είναι όμως δυνατόν με τη μία να ασχοληθούμε με όλα και με τις στρατηγικές και με τις, τη συνοχή των πολιτικών και την αποτελεσματικότητά τους και την αποτελεσματικότητα του φορολογικού ε, συστήματος κλπ. Αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει να κάνουμε συζήτηση σχετικά με το ποια είναι η αποτελεσματικότητά μας όσον αφορά την αναπτυξιακή βοήθεια. Αυτό σημαίνει ότι δεν χρειάζεται ε, να υπάρξει ευθυγράμμιση όλων των φορέων και εμπλεκομένων. Ε, όχι βέβαια και είναι γεγονός ότι ο κατακριματισμός δεν έχει δώσει καλά αποτελέσματα. Ναι, ε, αλλά σε πάρα πολλές περιπτώσεις ε, ε, προσπαθούμε να έχουμε μία πιο συνολική προσέγγιση με την κοινωνία των πολιτών, με την κεντρική κυβέρνηση και αυτό μπορεί από μόνο του να οδηγήσει σε κατακαιρματισμό. Ναι, υπάρχουν πολλά άλλα ζητήματα τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπιστούν έτσι ώστε να επιτευχθούν οι αναπτυξιακοί στόχοι, αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ένα συνολικό πλαίσιο συνεκτικό όσον αφορά τα κύρια κυβέρματα, τις προκλήσεις ε, και τις πιο οξύες ε, προκλήσεις. Ε, η Σουζάν θα μιλήσει για τον ρόλο της κοινωνίας των πολιτών. Ο χώρος που πρέπει να δοθεί στην κοινωνία των πολιτών ως βασικό πρωταγωνιστή μειώνεται σε πολλές περιπτώσεις και αυτό είναι πρόβλημα. Αυτό που θέλουμε εμείς είναι στα πλαίσια του ε, διαλόγου για, την, ε, ε, για τους πρωταγωνιστές του, του, του διαλόγου και στα πλαίσια του διαλόγου για την για την αποτελεσματικότητα της ανάπτυξης να συμπεριληφθεί και η κοινωνία των πολιτών. Αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς δεν θέλουμε ή δεν έχει λόγο ή ρόλο η κοινωνία των πολιτών σε άλλους τομείς. Απλώς θα πρέπει να βρεθούν ε, τα στοιχεία αυτά τα οποία είναι πιο σημαντικά. Δεν θα προσπαθήσω να απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις. Νομίζω ότι πολύ μεταξύ μόνο αναφέρατε ότι ε, ε, ε, ένα από τα building blocks ήταν αυτές οι ευάλωτες χώρες, fragile states, και γνωρίζετε ίσως ότι έχει δημιουργηθεί μια πλατφόρμα που αφορά τις ε, χώρες ε, ε, οι οποίες είναι πιο ευαίσθητες, οι οποίες αντιμετωπίζουν συγκρούσεις, να φέρουν σε επαφή λοιπόν μέσω της πλατφόρμας αυτής τις χώρες αυτές με τις χώρες της αναπτυξιακής βοήθειας. Υπάρχουν, έχουμε προχωρήσει στο θέμα της πλατφόρμας αυτής. Μπορώ να σας δώσω και κάποια στοιχεία για τον τρόπο με τον οποίο να διευθύνσετε Διάλογος προχωρήσει προχωράει. Επίσης θα ήθελα να απαντήσω στο κατά πόσον και πώς μπορούμε να είμαστε προβλέψιμοι ε, και πώς είναι δυνατόν αυτό ε, να το συνδυάσουμε με την ευελιξία. Καταρχήν το αν αυτές οι διέννησεις είναι αντιφατικές μεταξύ τους, προβλεψιμότητα και ευελιξία. Ξέρετε πως ε, ένα από τα διδάγματα που είχαμε τα τελευταία, αποκομίσει τα τελευταία χρόνια είναι πως θα πρέπει να είναι μακροπρόθεσμο το θεματολόγιο και όχι βραχυπρόθεσμο. Δεν μπορούμε να φέρουμε αυτή την αλλαγή σε τρία ή πέντε χρόνια. Οπότε είναι ανάγκη και νομίζω ότι σε αυτό συμφωνούν όλοι να έχουμε μακροπρόθεσμο όραμα, στρατηγική και στράτευση. Αυτό δεν σημαίνει πως θα πρέπει να χάσουμε και την ευελιξία μας να αντιμετωπίζουμε επίγουσες καταστάσεις, κρίσιμες καταστάσεις, για παράδειγμα το προσφυγικό το οποίο δεν ήταν τμήμα της μακροπρόθεσμου θεματολογίου όταν εμφανίστηκε. Όμως θα πρέπει όσοι λαμβάνουν αποφάσει και οι κυβερνήσεις εκτός από το μακροπρόθεσμο όραμα να μπορούν να προσφέρουν και μια απόκριση στις ε, προκλήσεις που παρουσιάζονται. Και τέλος, ναι, έχουμε προκλήσεις σε κρατικό επίπεδο και μας είπατε πως θα πρέπει να έχουμε περισσότερη στόχευση στην εφαρμογή ανακράτος. Πρέπει να σας πω πως αυτό γίνεται κάθε δύο χρόνια ε, σε σφαιρικό επίπεδο, αλλά συνέχεια σε κρατικό επίπεδο γίνεται η παρακολούθηση. Έχουμε σε οκτώ χώρες αυτή τη στιγμή μηχανισμούς εποπτείας για το κατά πόσο είναι αποτελεσματική αναπτυξιακή βοήθεια. Και είναι στην εφαρμογή ανακράτος ε, που βρίσκουμε τα επιχειρήματα για να χρησιμοποιήσουμε στην σφαιρική αξιολόγηση που γίνεται. Άρα λοιπόν η συμμετοχή της ε, κοινωνίας των πολιτών γίνεται και σε κρατικό επίπεδο. Ο ιδιωτικό κλάδος ε, εμπλέκεται σε ε, κρατικό επίπεδο. Αυτά συμβαίνουν. Όχι ότι δεν έχουμε προκλήσεις, είναι ένας χώρος στον οποίο ενδεχομένω θα χάσουμε το δυναμικό μας, γιατί έχουμε πετύχει κάποιους στόχους, θα πρέπει να τους διατηρήσουμε, θα πρέπει να τους προωθήσουμε, αλλά η αναπτυξιακή βοήθεια έχει αναλάβει την υποχρέωση αυτή. Αν χάσουμε τη δυνατότητα της εποπτείας του να τα φέρνουμε μπροστά σας και να σας λέμε εκεί δεν πήγαμε καλά και πώς μπορούμε να ξεπεράσουμε τα προβλήματα, τότε θα έχουμε πρόβλημα. Και αυτό πρέπει να διαπραγματευτούμε στο Ναϊρόμπι. Θα πρέπει αυτή η δέσμευση να συνεχίσει να υπάρχει, έτσι ώστε τα στοιχεία και η παρακολούθηση να είναι διαθέσιμα και θα είναι και διαθέσιμα τις επόμενες εβδομάδες για να συνεχίσει η συζήτηση που κάνουμε. Ευχαριστώ πολύ, Σουζάνα. Σας ευχαριστώ. Χαίρομαι που η έκθεση για την παρακολούθηση ε, θα φτάσει στα χέρια μας σύντομα, έτσι ώστε να δούμε τι θα γίνει σε επίπεδο Συμβουλίου και Κοινοβουλίου και να παρουσιάσουμε και συγκεκριμένες προτάσεις και δεσμεύσεις. Νομίζω πως είμαστε λίγος πολύ στην ίδια στο ίδιο μήκο κύματο με τι δικέ σα προτάσει και έχουμε και ένα πολύ καλό παράδειγμα που είναι αυτό που συναντάμε επί τόπου. Θα ήθελα να υπενθυμίσω το θέμα της ε, προβλεψιμότητας. Ένα θέμα πολύ ενδιαφέρον, γιατί όπως όλοι θυμόσαστε, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο πιο προβλέψιμος ε, δωρητής. Ο προϋπολογισμός μας καλύπτει μια περίοδο 7 ετών. Κανείς άλλος δεν έχει κάτι αντίστοιχο. Και έχουμε και δεσμεύσεις. Δεσμεύσεις από το 2001 ε, που έπρεπε να έχουμε πετύχει μέχρι το 2015. Και ξαφνικά Είπαμε το κονσένσους και κάθε χρόνο εξετάζαμε τα νούμερα για να δούμε πόση αναπτυξιακή βοήθεια ως ποσοστό της παγκόσμιας βοήθειας προσφέρει. Και κάθε βράδυ ποια είναι η σύστασή μας μέχρι το 2015 ήταν ένα επαναλαμβάνουμε τους στόχους, μέχρι το 2015 δεν τους πετύχαμε και γίναμε πιο εφευρετικοί. Και τώρα αυτό που προσπαθούμε να πετύχουμε είναι να φτάσουμε το 0,7% ε, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες του προπολογισμού ε, κάθε έτος. Το οποίο σημαίνει ότι έχουμε κα, ε, κάτι πολύ ασαφές. Είπαμε 0,7 μέχρι το 2030. Μα αυτό είναι εξαιρετικά αργά. Και αυτό είναι το δίδαγμα του προηγούμενου 1,7%. Χρειάζεται στόχο. Ένα στόχος που θα έχει μια προθεσμία πιο σύντομη από το 2030 και να σας υπενθυμίσω πως η βοήθεια, η αναπτυξιακή, είναι ε, ένας από τους ασφαλείς πόρους. Ε, αν δείτε, ακόμα και κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής ε, κρίσης, οι εκροές ε, βοήθειας δεν εξαφανίστηκαν. Οπότε στις χώρες επί τόπου, παρόλο την κρίση, συνέχισαν να φτάνουν αυτά τα κονδύλια με σκοπό την εξάλληψη της φτώχειας. Και βέβαια δεν έχει να κάνει μόνο με τους αριθμούς. Έχει να κάνει με την αποτελεσματικότητα αυτών των αριθμών. Έχουμε τις δεσμεύσεις, έχουμε τις αρχές, ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Δεν χρειάζεται να επανεφεύρουμε τον τροχό. Δεν χρειάζεται να κοιτάμε το ποτήρι που είναι μισογεμάτο ή που είναι μισοάδιο. Όχι, πρέπει το ποτήρι να το γεμίσουμε το συντομότερο δυνατόν. Γιατί διαφορετικά ο κόσμος αλλάζει. Δεν είναι μόνο το προσφυγικό, έχουμε και άλλες προκλήσεις που πολύ σύντομα θα χρειαστεί να αντιμετωπίσουμε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ και σας ευχαριστώ που μας υπενθυμίσατε που παρόλο που τρέχουν αυτή τη στιγμή κάποια προβλήματα, η κατάσταση γενικά έχει βελτιωθεί. Έχουμε φύγει από το επίπεδο των έργων, από τη συνδεδεμένη βοήθεια και τα τελευταία 15-20 χρόνια είδαμε να έχει αλλάξει το θεματολόγιο, αλλά χρειάζεται χρόνος. Ακόμα και στις δικές μας χώρες, στην Ευρώπη, χρειάζεται χρόνος. Ε, βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή ε, στην... Ε, σε περιοχές όπου 30 χρόνια μετά την ε, εξάλληψη της ανθρακοβιομηχανίας ακόμα έχουμε κοινωνικά προβλήματα. Οπότε αυτό θα πρέπει να το θυμόμαστε. Μπορούμε να ευχαριστήσουμε λοιπόν τους δύο μιλήτρες. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε. Ο κύριος Πρέντα χρειάστηκε να φύγει. Έχει μια άλλη συνάντηση. Θα παρουσιάσει την ε, έκθεσή του για να την ε, παρουσιάσει στις 10 Οκτωβρίου τροπολογίες μέχρι τις 17 Οκτωβρίου για να ψηφίσουμε την έκθεση το Νοέμβριο και να εγκριθεί πριν τον Ναϊρόμπι. Ευχαριστώ πολύ. Περνάμε λοιπόν και στο επόμενο και τελευταίο σημείο τη ημερήσια διάταξη, που είναι η προώθηση τη ισότητα των φύλων στην ψυχική υγεία και την κλινική έρευνα. Είναι μια γνωμοδότηση από την Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών Ισότητα των Φύλων. Κύριε Σεβαστιά, είστε ο εισηγητή. Καλημέρα σας. Κυρία Πρόεδρε, ξέρετε πως πρόκειται για μια γνωμοδότηση, για μια έκθεση που έρχεται από την Επιτροπή Δικαιωμάτων Γυναικών και Ισότητας των Φύλων, όπου και εγώ συμμετέχω, οπότε είπε σε άμεση επαφή με την εισηγήτρια εκεί. Υπάρχει μια συντηρητική, παραδοσιακή, πατριαρχική ε, αντίληψη των κοινωνιών μας ε, που δεν χτίζει μόνο τείχους στην προσπάθεια πρόσβαση των γυναικών στην ισότητα, όχι μόνο στον ιδιωτικό χώρο αλλά και στο δημόσιο χώρο, αλλά έχει κατακλείσει όλο μας την κοινωνία και ε, την επιστήμη και την ιατρική έρευνα και την ιατρικές θεραπείες που βασίζονται στα όσα επηρεάζουν τους άνδρες χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τις βιολογικές και φυσιολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών. Η έκθεση αυτή έχει ως σκοπό να ξεπεράσει αυτές τις δυσκολίες, να λάβουν μέτρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην έκθεση που έχει η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών μας έδωσε την ευκαιρία μέσω της δική μας γνωμοδότησης να υπενθυμίσουμε Ποιε υποχρεώσεις έχει αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, στην, ε, στα θέματα συνεργασία και ανάπτυξης ε, σε αυτούς εδώ τους κλάδους. η ομάδα μας παρουσιάζει μια σύντομη γνωμοδότηση περιορισμένης κλίμακας όπου τονίζουμε κάποια σημεία. Τα δύο πρώτα σημεία μας υπενθυμίζουν τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την καθολική ε, διάσταση και ζητά από τις χώρες να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα να ξεπεραστούν οι διακρίσεις που βασίζονται στο φύλλο, όχι μόνο σε θέματα υγείας, αλλά και στην ιατρική έρευνα που γίνεται. Και κατόπιν έχουμε τρία σημεία τα οποία είναι ουσιαστικά και στα οποία πιστεύουμε πως θα πρέπει εμείς να στείλουμε ένα απερίφραστο μήνυμα στα ευρωπαϊκά όργανα. Καταρχήν, με λύπηση διαπιστώνουμε πως αυτή η ευρωπαϊκή στρατηγική δεν λαμβάνει υπόψη την παγκόσμια πολιτική για θέματα υγεία. Υπάρχει μια έλλειψη δέσμευσης για τις αρχές αυτές, για την υγειονομική περίθαλψη, ε, παρόλο που εμεί έχουμε ζητήσει και στην στρατηγική για την καινοτομία και την έρευνα τη Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχουν ληφθεί δεόντως υπόψη. Δεύτερον, σημειώνουμε με ανησυχία ότι παρόλο που στηρίζουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση την έρευνα έτσι ώστε να ξεπεράσουμε την έλλειψη φαρμάκων ε, και θεραπείων για αυτές τις ξεχασμένες ή αγνοημένες ε, ασθένειες οι οποίες συνδέονται με τη φτώχεια και επηρεάζουν τα πιο φτωχά κράτη, τα κράτη που είναι ε, στην πορεία της ανάπτυξης έρευνες δεν γίνονται, κλινικές δοκιμές δεν γίνονται και προσφέρει βοήθεια η Ευρωπαϊκή Ένωση έτσι ώστε να ερευνώνται αυτές οι ασθένειες αλλά δυστυχώς δεν φτάνουν τα κονδύλια αυτά έτσι ώστε οι ιατρικέ έρευνες να προσφέρουν πραγματικά φάρμακα τα οποία θα είναι διαθέσιμα διαθέσιμα και σε αυτούς τους πληθυσμούς. Αυτό θέλουμε να διορθωθεί. Επίσης, υπάρχει ένα ιδιαίτερα δύσκολο θέμα που είναι η μετεγκατάσταση των ε, δοκιμών φαρμάκων. Οι, τα μεγάλα, οι μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες έχουν μετατοπίσει τις κλινικές δοκιμές. Είναι ευρωπαϊκές εταιρείες και οι δοκιμές γίνονται στην Αφρική. Είναι γνωστό γιατί είχαμε πολλές εκθέσεις και μάλιστα και μια πολύ γνωστή ταινία για το γεγονός πως ο πληθυσμός ε, στις ε, χώρες που είναι πιο φτωχές πολλές φορές μπαίνει ε, σε αυτές τις κλινικές δοκιμές γιατί είναι η μοναδική δυνατότητα που έχουν να λάβουν κάποιο είδους θεραπεία για τις ασθένειες αυτές από τις οποίες υποφέρουν και πολλές φορές ε, δεν ερευνούνται επαρκώς και πολλές φορές έχουμε ε, κατάφορες παραβιάσει θεμελιωδών δικαιωμάτων εδώ, όπως οι ασθενεί ε, που παίρνουν μέρος σε αυτές τις έρευνες δεν προστατεύονται, δεν ε, ενημερώνονται και πολλές φορές έχουν και κάποιες επιπτώσεις από αυτές τις δοκιμές φαρμάκων που δεν αναλαμβάνονται μετά από τις φαρμακευτικές που κάνουν τη δοκιμή και τελικά λειτουργούν ω απλά πειραματόζωα νομίζω ότι θα πρέπει να προστατεύονται πιο πολύ τα δικαιώματά τους. Αυτές είναι οι γενικές γραμμές ε, που θα ακολουθήσουμε. Πάντα έχουμε πρόβλημα χώρου και χρόνου, αλλά νομίζω πως εάν θέλετε να συνεισφέρετε, αυτό το μόνο που θα κάνει είναι να εμπλουτίσει το κείμενό μας και η σχέση μας με την Επιτροπή Δικαιωμάτων Γυναικών είναι ρέει πιο εύκολα τώρα που είμαι και εγώ μέλος και θα ήθελα να ζητήσουμε όλοι μαζί η Ευρωπαϊκή Ένωση να ε, συμμορφωθεί με τα όσα έχει ήδη εγκρίνει στις συνθήκες της. Ευχαριστώ πολύ. Έχω τρεις ομιλητές που έχουν ζητήσει το λόγο. Η κυρία Ζαμπόρσκα, η Μαρία Αλμπιόρ και η κυρία Ποιος άλλος θέλει το λόγο. Γιατί ξέρω πως δεν έχουμε πολύ χρόνο. Αυτοί οι τρεις ομιλητές έχουν το λόγο. Και ο κύριο παρακαλώ. Άννα Ζαμπόρσκα. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για το γεγονός ότι ετοιμάσατε αυτή την ε, γνωμοδότηση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω λοιπόν τον εισηγητή και να σας υπενθυμίσω πως από τότε που είμαι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, από το 2004, η Επιτροπή Γυναικών ξεκίνησε με μια πρώτη έκθεση για την περίθαλψη και τα θέματα φύλου που σχετίζονται με την παροχή ε, περίθαλψης. Η πρώτη έκθεση μάλιστα παρουσιάστηκε το 2005. Αυτό που μόλις ανέφερε λοιπόν ο συνάδελφός μας ο συγητής, όλες οι επιφυλάξεις που έχουμε για την παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στις άνδρες, στις γυναίκες και στις διαφορές που υπάρχουν, έχουν ήδη περιγραφεί στην έκθεση αυτή και το πρώτο μου σχόλιο είναι πως ίσως θα έπρεπε να ξαναδούμε αυτές τις εκθέσεις, οι οποίες, επαναλαμβάνω, είχαν ε, παρουσιαστεί από μεμονωμένες επιτροπές στο παρελθόν για να αξιολογήσουμε ποιες ήταν και οι εξελίξεις τα τελευταία 15 χρόνια. Κυρίως όσον αφορά τη γνωμοδότηση ε, που παρουσιάζει ο εισηγητής, να τον συγχαρώ θεωρώ πως ε, έχει πραγματικά κατανοήσει και περιγράψει τα σημαντικά σημεία, κυρίως για την ψυχική υγεία των γυναικών και για την αναπτυξιακή πολιτική στα σχετικά θέματα. Πιστεύω πως ε, υπάρχει χώρος στην ε, αναπτυξιακή πολιτική για να συμπεριλάβουμε και τα θέματα ψυχικής υγείας και ψυχικών διαταραχών. Δεν θέλω να υπονοήσω πως στις αναπτυγμένες χώρες όπου υπάρχει διαφορετικό επίπεδο άγχος, δεν έχουμε ψυχικές διαταραχές στις άνδρες και στις γυναίκες, αλλά στις αναπτυσσόμενες χώρες η κατάσταση είναι πολύ συγκεκριμένη. Γιατί? γιατί έχουν το μακροπρόθεσμο άγχος που προκαλεί η φτώχεια, για παράδειγμα. Οι σειράξει, οι πόλεμοι και που επηρεάζουν κατά κύριο λόγο τις γυναίκες. Εκτός λοιπόν αυτού του εξωγενείς αρνητικούς ε, παράγοντες, έχουμε γυναίκες που πρέπει να μεγαλώσουν την οικογένειά τους και επηρεάζονται πάρα πολύ από τις αρνητικές συνέπειες των πολέμων, των σειράξεων, της πείνας, της φτώχειας. Και για το λόγο αυτό, οι γυναίκες αυτές πολύ δύσκολα υπό αυτές τις συνθήκες καταφέρουν να λάβουν την κατάλληλη θεραπεία, γιατί όπως σας είπα και προηγουμένως, η κατάστασή τους και η ψυχική τους υγεία τις οδηγούν σε έναν κύκλο αδυσόπιτο και για τον λόγο αυτό πιστεύω ότι χρειάζεται περισσότερη συμβολή ε, των ευρωπαϊκών θεσμών έτσι ώστε να λάβουμε υπόψη και το θέμα της ψυχικής υγείας των γυναικών στις ε, χώρες στις οποίες πηγαίνει η αναπτυξιακή μας βοήθεια πώς εξασφαλίζοντας πως η αναπτυξιακή μας πολιτική ε, θα λάβει κάποια μέτρα έτσι ώστε να είναι πιο πετυχημένη και οι γυναίκες στα κράτη αυτά θα προστατεύονται μέσω αυτών των οντικών μας πολιτικών. Πιστεύω πως ο συνάδελφος τόνισε τα πιο σημαντικά σημεία και κυρίως για το σημείο 3 όπου αναφέρεται στους εξωτερικούς παράγοντες που επηρεάζουν ε, ε, τις γυναίκες τα είπε πολύ σωστά ο κύριος Τσούλικα, σας παρακαλώ. Ε, πιστεύω πως έχει σχεδιαστεί πολύ σωστά αυτή η γνωμοδότηση. Θα συνεργαστούμε με τον εισηγητή. Πιστεύω, αγαπητοί συνάδελφοι, πως όλοι θα συμφωνήσουμε στο εξής θα πρέπει με στεναρό τρόπο να καταπολεμήσουμε τις διακρίσεις και να προωθήσουμε την ισότητα των φίλων σε όλους τους χώρους. Οι γυναίκες αντιμετωπίζουν τα δικά τους θέματα υγείας. Και όπως γνωρίζουμε, είναι και στις αναπτυσσόμενες χώρες πιο ευάλωτες. Εάν χρειάζεται οι υπηρεσίες υγείας να αντιμετωπίσουν τις ανάγκες γυναικών και ανδρών, θα πρέπει ε, τα ιδιάζοντας χαρακτηριστικά να ληφθούνται όντως υπόψη ε, στη χάραξη στρατηγικής και θα πρέπει να δούμε πώς η συμπεριφορά τους, η οικογενική τους κατάσταση, η θέση τους στην κοινωνία επηρεάζει το κατά πόσο έχουν πρόσβαση, ισότιμη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας. Απευθύνω λοιπόν μια πρόσκληση στις χώρες, ε, στις κυβερνήσει των ε, χωρών σε ανάπτυξη να εντάξουν το θέμα αυτό στην ε, πολιτική τους, στην πολιτική υγεία και να έχουν και το θέμα της ψυχικής υγείας των γυναικών ε, στα στις προσπάθειες που θα κάνουν και με χαρά θα συνεχίσουν να συνεργάζομαι με τον εισηγητή στα θέματα αυτά. Η κυρία Αλμπιόλ. Ευχαριστώ. Θέλω απλώς να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την εργασία του και την πρότασή του. Συμφωνώ απόλυτα με τα θέματα που θέτει. Σίγουρα υπάρχουν ανισότητες, διακρίσεις ε, για λόγους φύλου στην έρευνα, παντού στον κόσμο και στην Ευρώπη <clears throat> και φυσικά και στις ε, φτωχές χώρες που είναι θέμα αρμοδιότητας της Επιτροπής μας. Ευχαριστώ τον εισηγητή γιατί αναφέρεται σε αυτές τις συνήθειες των ε, πολυεθνικών που επιτείνουν αυτήν την ε, ανισότητα μέσω των ε, κλινικών δοκιμών και ότι πρέπει να υπάρχει δημόσια παροχή περίθαλψης που είναι ουσιώδης αν θέλουμε να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα. Εμείς η Ευρωπαϊκή Αριστερά θα υποβάλουμε κάποιες τροπολογίες αλλά απλώς για να συμπληρώσουμε αυτά τα οποία έχει ήδη παρουσιάσει ο εισηγητής. Ε, θέλουμε να υπάρξει περισσότερη προσοχή για την πρόληψη, να μην στιγματίζονται και να συμπεριληφθούν και οι κοινότητες LGBTI, αλλά όπως σας είπα γενικά συμμεριζόμεθα την αντιμετώπιση του και τα θέματα στο οποία εστιάζει. Ευχαριστώ όλοι και Σαρλ Γκερένς, τελευταίος αλλά όχι λιγότερο σημαντικός. Ευχαριστώ και εγώ τον εισηγητή. Το αποτέλεσμα της εργασίας του είναι νομίζω ιδιαίτερα θετικό. Κυρίως με απασχολεί το σημείο 3 όπου, όπως λέει και ο συγητής, ε, εκφράζει τη λύπη του για το ότι δεν υπάρχει κανένας μηχανισμός ε, που να φροντίζει με υποχρεωτικό τρόπο ε, που να επιβάλλει με υποχρεωτικό τρόπο την παροχή φαρμάκων με προσβάσιμες τιμές. Το θέμα αυτό ήταν ε, μία αιτιολογική σκέψη της έκθεσής μου για την, για την ε, έμπολα. Είχαμε ασχοληθεί με το θέμα, τι θα κάνουμε εάν η αγορά ή οι φάρμακοβιομηχανίες δεν παράγουν προϊόντα για την αντιμετώπιση σπανίων ασθενειών ή για το πώς θα χορηγηθούν φάρμακα για, σε ασθενείς που δεν έχουν τα μέσα για να τα αγοράσουν. Και θέλαμε η Επιτροπή ΕΝΒΙ και η δική μας να κάνει μια έκθεση για το θέμα αυτό. Ελπίζω λοιπόν ο εισηγητής ε, να λάβει υπόψη το θέμα αυτό. Νομίζω ότι ε, μία σύντομη τροπολογία θα μπορούσε να συμπεριληφθεί. Χαίρομαι που η συζήτηση αυτή γίνεται με ηρεμία και αυτό οφείλεται στο ότι δεν υπάρχουν φαλοκράτες μεταξύ μας. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Στο 13 θα συζητήσουμε την πρόσβαση στα φάρμακα, γνωμοδότηση για την ένβη. Σήμερα το απόγευμα. Ωραία. Ο κύριος Μπαστιά θέλει να προσθέσει τίποτα. <clears throat> ναι, ευχαριστώ και εγώ για τα σχόλια από όλους μου τους συναδέλφους. Το γεγονό ότι όλοι συμφωνούμε καθιστά προφανές ότι είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα που πρέπει οπωσδήποτε να αντιμετωπιστεί. Φυσικά δέχομαι αυτό που πρότεινε ο κ. Γκέρενς. Ελπίζω λοιπόν ότι θα μου υποβάλει την τροπολογία και φυσικά θα την ε, εντάξω. Και επίση πολύ ενδιαφέροντα αυτά που λέει συνάδελφος Αλμπιόλ που είπε ότι πρέπει μέσω τροπολογιών να ε, τονίσουμε περισσότερο την πρόληψη ναι, ναι, βεβαίως. Ε, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στην έκθεση. Θα την εμπλούτιζε ιδιαίτερα. Και για τη Σάνφο Ζαμπόρσκα. Βεβαίω και δέχομαι αυτό που μας είπε. Να δούμε αν η έκθεση στην οποία αναφέρθηκε το 2005, η κατάσταση τότε, ε, έχει αλλάξει έκτοτε. Και δεν νομίζω ότι έχουν αλλάξει πολλά. Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον λοιπόν να κάνουμε αυτή τη σύγκριση. Αναμένω λοιπόν αυτές τις ε, συμπληρώσεις γιατί νομίζω ότι θα είναι πολύ σαφής και πολύ κατηγορηματική η γνωμοδότησή μου. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι βασικό είναι να είμαστε σύντομοι γιατί αλλιώ μπορεί να επηρεάσει, γιατί με αυτόν τον τρόπο θα επηρεάσει περισσότερο την ε, Επιτροπή ε, Γυναικών. Όσο λιγότερε τροπολογίε υποβάλλουμε, τόσο το καλύτερο. 8 Σεπτεμβρίου 12 η προθεσμία, η ψηφοφορία. στι 8 Νοεμβρίου ευχαριστώ τον κύριο Σεβαστιά Οπότε λίγη συνεδρίασή μας σήμερα το πρωί. Συνάδελφοι, στι 3 έχουμε πολλές ψηφοφορίε, Παρακαλώ, μην ξεχάσετε τις κάρτες σας. Τα λέμε τότε.